Συνάδελφοι, λέω να αρχίσουμε. Δεν έχουν έρθει ακόμη όλοι και όλες, αλλά έχουμε φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Γι' αυτό ας μην χάσουμε πολύ χρόνο. Ίσως είδατε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα τώρα να προτείνω μερικές, όχι αλλαγές, όχι αλλαγές, αλλά αποσαφηνήσεις για τη σειρά με την οποία θα εξετάσουμε τα διάφορα θέματα. Θα αρχίσουμε από την έκθεση Γκάγερ γιατί ένα σημαντικό διεθνές τηλεοπτικό κανάλι ήρθε από τώρα και θα αρχίσουμε από εκείνο το θέμα μετά έκθεση Βαρβάρας Ματέρα αν είναι εδώ είναι ναι ναι αμέσως μετά τον κύριο Γκάγερ θα ακούσουμε τη δική σας έκθεση όπως ζητήσατε και να φροντίσουμε το θέμα του πολιετούς ε, δημοσιονομικού προγράμματος πριν τις 10 και 40 να το τελειώσουμε γιατί θα φύγει τότε ο Μπέγκε και ο Ράιμερ. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις λοιπόν αυτές οι αλλαγές, ε, όπως είπα δεν ήταν αλλαγές αλλά θα ήθελα τώρα να εκφράσω τη χαρά μου διότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της γυναίκας και των γυναικών Χαιρετίζω όλες τις γυναίκες που μας τιμούν με την παρουσία τους για την αποτελεσματικότητά τους, τα ικανότητες τους και το... την ομορφιά τους. Συγχαίρω επίσης και τη συνεργάτιδές μας. Τουλάχιστον τα δίσεκτα έτη καλό είναι να εορτάζομαι τις γυναίκες. Λοιπόν, ανακοινώσει του Πρόεδρου. Επειδή δεν έχουν ακουστεί αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό της Συρίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από τη δάνεια της ΕΟΤΕ εγκρίνεται η πρόταση. Απ' την άλλη σας πληροφορώ ότι οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου αρχίζουν ένα πείραμα στα πλαίσια των εργασιών μιας ειδική επιτροπής για την κατάργηση του χαρτιού μέσω των διαφόρων μεθόδων ήτα, ηλεκτρονικών δηλαδή. Ως Επιτροπή Προϋπολογισμών, διότι η πρόταση αυτή αφορά όλες τις επιτροπές του Κοινοβουλίου, θα φροντίσουμε να μοιράσουμε 5-6 iPad και εδώ και μερικές εβδομάδες θα γίνει αυτό το πείραμα οι συνάδελφοι να χρησιμοποιούν το iPad εφόσον υποσχεθούν να μην ξαναχρησιμοποιήσουν χάρτην. Ακούω υποψηφιότητες και θα επιλέξω αν υπάρξουν πολλές υποψηφιότητες παραπάνω από τα διαθέσιμα iPad θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τέλος, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι κατά τη τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών και συντονιστριών συμφωνήσαμε να γίνουν ορισμένοι ορισμοί. Ashworth ορίστηκε εξ ονόματος των συντηρητικών εισηγητής για την καταπολέμηση των ατών και για τα προγράμματα Φίσκας και Ηρακλής 3 καθώς και Περικλής. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Στατιστικής. Η Συθωνία ορίστηκε εισηγήτρια για το πρόγραμμα Έρασμος για όλους. Και ο ορίστηκε για το ΙΠΑ. ΙΠΑ. Εν μεταξύ ο συνάδελφο Σαμπάντ έφυγε από την Επιτροπή Προπολογισμών, πράγμα για το οποίο λυπόμαστε ιδιαίτερα, αλλά αντικαταστάθηκε από τον κύριο Κοσλόφσκι, που νομίζω ήρθε και όλα σήμερα. Όχι, δεν ήρθε ακόμα, δεν ήρθε ακόμα, αλλά θα έρθει. Ο κύριος Κοσλόφσκι λοιπόν που είναι των συντηρητικών, όχι του ΕΛΚ είναι του ΕΛΚ, του και ανέλαβε και τα θέματα του προκατόχου του. Ναι, τέλος πάντων δεν ξύπνησα πολύ φρέσκος, αλλά τι να γίνει. Και η Μαρία Καρβάλιο... Le point 3. Αντικαταστάθηκε και αυτή. Τρία. Τα πρακτικά για την προηγούμενη συνεδρίασή μας 6 Φεβρουαρίου σύμφωνα με τη Ιωθώτα αν δεν ακουστούν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος τη συνεδρίας θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκουρηθεί. Και πάμε τώρα αμέσω χωρίς καθυστέρηση στο σημείο 10 που είναι, που είναι λέγω το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή κύριο Γκάιερ. Ähm, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που έχετε προτάξει τη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σήμερα το πρωί ως αρμόδιοι για τον προϋπολογισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς δίνουμε μια γρομοδότηση στην Επιτροπή Απασχόλησης. Το πλαίσιο όλων αυτών είναι η νέα οδηγία για το κοινωνικό ταμείο στην επόμενη περίοδο δημοσιονομικού σχεδιασμού. Έχουμε βέβαια περίπου 30 εκατομμύρια ανέργων και 110 εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι απειλούνται από την ένδυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει το καλύτερο εργαλείο της για την αντιμετώπιση της ανεργίας που είναι το κοινωνικό ταμείο Περαιτέρω, <clears throat> χρειάζεται να αναπτύξουμε και στρατηγικές για καλύτερη αντιμετώπιση της ανεργίας. Θα πρέπει να αυξήσουμε την κινητικότητα των εργαζομένων μέσα στην Ευρώπη και να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι καλύτερες οι συνθήκε που θα επιτρέπουν την κοινωνική τους ενσωμάτωση. <clears throat> Μας προτείνει τέσσερις θεματικούς στόχους η Κομισιόν. Καταρχήν η υποστήριξη της κοινοτικότητος, η εκπαίδευση, κατάρτιση και διαβίου ε, εκπαίδευση, κοινωνική ενσωμάτωση και τέλος η πιο αποτελεσματική δημόσια δίκηση και η αύξηση των ικανοτήτων. Αυτά είναι θέματα τα οποία το τελευταίο θέμα δεν συμπίπτει απόλυτα με αυτά τα οποία έχει να κάνει το κοινωνικό ταμείο, αλλά εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι γίνεται σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων και νομίζω ότι εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα θετικό παράδειγμα σε ό,τι αφορά τα ασφάλματα και τις, ε, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην ε, εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ξέρουμε ότι για πάρα πολλές περιοχές η χρήση του Κοινωνικού Ταμείου είναι ένας πραγματικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτών των περιοχών. Λέγεται ότι αυτοί οι τέσσερις στόχοι θα πρέπει να υλοποιηθούν ως προτεραιότητες, αλλά πάντα με τη συνεργασία των περιφερειών. Θα πρέπει να δούμε ποιοι στόχοι είναι οι πιο σημαντικοί για κάθε συγκεκριμένη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κομισιόν και των περιφερειών της Ευρώπης. Η Κομισιόν θέλει ούτως ή άλλως το 20% τουλάχιστον των πόρων του Κοινωνικού Ταμείου να έχει σε στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση <clears throat> και επί τη βάση των τριών επιπέδων που προβλέπονται για την πολιτική συνοχή θα πρέπει οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές να έχουν μια επιδότηση τουλάχιστον 25%, 40% στη μεσαία περιοχή και 25% για το υψηλότερο επίπεδο και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει και κάποια έλλειψη <clears throat> συνένεσης μεταξύ των επιτροπών που έχουν να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά, γιατί η Επιτροπή Απασχόληση θεωρεί θετικά αυτά τα ποσοστά, η Επιτροπή Περιφερειακών θεμάτων θεωρεί ότι δεν συμφωνεί γιατί αναρωτιέται αν θα πρέπει οι πιο ανεπτυγμένες περιοχές να καταλάβουν παρόλα αυτά 25% του κοινωνικού ταμείου. Μήπω οι περιοχές οι οποίες έχουν επιτύχει την πλήρη απασχόληση να αφήσουν τα κονδύλια τους για να χρησιμοποιηθούν σε φτωχότερες περιοχές. Αυτά είναι η απόψη της Επιτροπής Περιφερειακών Θεμάτων. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαμε από τη μία πλευρά <clears throat> να περιοριστούμε στο να εξετάσουμε τα άρθρα 13, 14, 15 που αφορούν την οικονομική διαχείριση και να παραμείνουμε έτσι πιστοί στη δική μας εντολή ως χνομοδοτική Επιτροπή. Εγώ Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συζητήσουμε και να εξετάσουμε και την αποτελεσματικότητα των χρηματοδόσεων. Νομίζω ότι η Κομισιόν προτείνει να υπάρξουν καταβολές επίσης ποσών κατά αποκοπή, όταν βλέπει κανείς τα μικρά προγράμματα με την συμμετοχή ΜΚΟ, μικρών ΜΚΟ που βοηθούν ομάδες που χρειάζονται πραγματικά βοήθεια, ομάδες του πληθυσμού που είναι ευάλωτες, είναι πολύ καλό για τις μικρές αυτές ε, ΜΚΟ που κάνουν μικρά σχέδια, που εφαρμόζουν μικρά σχέδια, να τις χρηματοδοτούμε κατά αποκοπή και να τις απαλλάξουμε από το γραφειοκρατικό βάρος. <clears throat> Επίσης η πρόλαση της Κομισιόν περιλαμβάνει και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Κομισιόν προτείνει να υπάρξουν ε, διάφορες μορφές ταμείων, ε, υποστήριξη για κεφάλαια κινδύνου, για κοινοπραξίες κτλ. Εμείς έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά με τον εισηγητή επί της ουσίας, αλλά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα για το κατά πόσο αυτά τα εργαλεία είναι τα πρέποντα ή όχι. Μπορεί να υπάρξει βέβαια κάποια διαφορά απόψεων μεταξύ μας σε σχέση με την υποχρέωση εκθέσεων που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή αυτών των εργαλείων και τον απαραίτητο έλεγχο που πρέπει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Και από αυτή την άποψη, εάν δεν υπάρχει αυτό, δεν πρέπει να εφαρμοστούν αυτά τα εργαλεία. Η υπομορφή τώρα κατεξουσιοδότηση πράξης <clears throat> έχει υπάρξει κάποια ε, παραχώρηση ε, αρμοδιοτήτων στην Κομισιόν που είναι ανακλητή. Υπάρχει μια συγκεκριμένη προθεσμία για να παρέμβουμε όταν η Κομισιόν πάρει μια απόφαση η οποία δεν βρίσκει την σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά εμείς φυσικά και ως ε, αρχή επί του προϋπολογισμού θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω για το θέμα αυτό, για το κατά πόσο η Κομισιόν θα πρέπει να έχει πράγματι αυτό το δικαίωμα να δρά βάσει εξουσιοδοτήσεων. Θα ήταν ε, επίσης απαραίτητο να βγούμε από το στενό πλαίσιο του προϋπολογισμού και να έχουμε μια ευρύτερη αντιμετώπιση για τα θέματα του κοινωνικού ταμείου. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω και μια συζήτηση αν και κατά πόσον αυτά τα μέτρα είναι τα καταλληλότερα για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία στην Ευρώπη. Αλλά περαιτέρω έχουμε και το ερώτημα ποιοι στόχοι θα πρέπει να καλύπτονται από ποιο διαρδοτικό ταμείο. Λέει η Κομισιόν πρέπει να υπάρχει και συνέργεια μεταξύ των διαρδοτικών ταμείων. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα ήταν καλύτερο ανάμεσα στο κοινωνικό ταμείο και το νέο πρόγραμμα για την κινητικότητα και την καινοτομία που προετοιμάζεται μήπως θα ήταν καλύτερο να έχουμε χαράξει πιο σαφείς οριοθετικές γραμμές μεταξύ των δύο αυτών πηγών χρηματοδότησης, ώστε να έχουμε μια πιο σωστή στοχοθέτηση για τη χρήση των πόρων αυτών και <clears throat> επίσης για το αν το κοινωνικό ταμείο μπορεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούσε να υπάρξει μια συμβολή του Κοινωνικού Ταμείου. Ίσως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο φιδωλοί και να μην θεωρούμε ότι όλοι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποιον εφελαιόδη τρόπο μπορούν να υποστηριχθούν από το Κοινωνικό Ταμείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Έχουν ζητήσει δύο συνάδελφοι το λόγο. Πρώτος ο κύριος Σούριαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τις τελευταίες φράσεις του εισηγητή αλλά και με τα υπόλοιπα και με τα υπόλοιπα, τα προηγούμενα δηλαδή. Θα ήθελα απλώ να σχολιάσω σύντομα πώς βλέπουμε εμείς αυτά τα θέματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ταμείο που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και η ανεργία υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούμε σωστά τα κονδύλια αυτού του ταμείου ανταποκρίνεται στους στόχους του ή μήπως πρέπει να τους αλλάξουμε. Το κοινωνικό ταμείο, η ανεργία είναι θέματα που πρέπει να μας οδηγήσουν σε κάποιες σκέψεις. Ίσως υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια κτίδα φωτός ότι φέτος δηλαδή μπορεί να καταλήξουμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικότερα τα προτινόμενα στη στρατηγική 2020 που είναι ο κύριος μας στόχος και πρέπει να προσαρμόσουμε τη λειτουργία του Ταμείου και τον προϋπολογισμό στους στόχους αυτούς. γιατί δεν, έχουν, δεν υπάρχει ειδικό ταμείο για την πραγματοποίηση των στόχων 2020. Συμφωνώ με την Κομισιόν ότι πρέπει να πλησιάσουμε, να συγκλίνουμε τους προγραμματισμούς όλων των παρεμφερών ταμείων, την πολιτική συνοχής, περιφερειακή ανάπτυξη, όλα αυτά. Όλα αυτά λέγω είναι παρεμφερή και νομίζω ότι το Ταμείο Ανάπτυξης της Υπέθρου αποτελεί και αυτό το τμήμα αυτών των παρεμφερών ταμείων. Υπάρχουν τρεις επίτροποι που ασχολούνται με αυτά και νομίζω ότι αυτό δεν ευνοεί την καλύτερη δυνατή λειτουργία των ταμείων αφού έχουν περίπου τους ίδιους στόχους όλα. Υπάρχει πάντως κάποια ελπίδα γιατί η Κομισιόν επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου για να μπορέσει να μετρήσει σε ποιο βαθμό υπάρχει και ποια αποτελεσματικότητα στη χρήση των όλων αυτών των ταμείων. Έτσι θα μπορούσαμε ίσως να ανταποκριθούμε το πρόβλημα της ανεργίας με την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση αυτών των ταμείων να την καταπολεμήσουμε. Εμείς θα θέλαμε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης τους αν και βλέπουμε ότι υπάρχουν και ορισμένοι κίνδυνοι και δυσκολίες στην εποπτεία και τον έλεγχο. Πρέπει οι περιφέρειες να μας δίνουν περισσότερα στοιχεία. Ούτως ή άλλως έχουμε την εντύπωση ότι ακόμη και αν όλοι αν και όλοι μιλάνε για απλοποίηση της χρήσης των ταμείων, αυτή η απλοποίηση δεν υπάρχει ακόμα. Δεν τη βλέπουμε πουθενά. Επίσης έχουμε την εντύπωση ότι το διοικητικό άχθος αυξάνεται συνεχώς. Αυτή είναι η θέση του ΕΛΚ, κύριε Πρόεδρε, και νομίζω ότι όταν θα έχουμε την τελική έκθεση και αφού ακούσουμε τον εισηγητή, θα είμαστε ίσως σε θέση και να τον υποστηρίξουμε και να δούμε κατά πόσον θα μας ακούσει και η αρμόδια επί της ουσίας Κοινωνική Επιτροπή. Δεν μιλήσαμε ακόμη για αριθμούς γιατί δεν είναι ακόμη τελική Θα γίνουν πάντως οι απαραίτητες διορθώσεις εν καιρό το δέοντι. Ο κύριος auch. Θα προσπαθήσω και εγώ λιγάκι να μιλήσω στα γερμανικά. Για μένα το πρώτο στοιχείο είναι ότι αν δούμε τα αποτελέσματα της 1ης ε, Φεβρουαρίου τι βλέπουμε βλέπουμε να υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των χωρών που είναι καλές σε απορρόφηση των πόρων του Κοινωνικού Ταμείου και τις άλλες. 63% είναι το ρεκόρ σε απορρόφηση, 19% είναι το χαμηλότερο επίπεδο. Υπάρχουν και χώρες μέσα στη ζώνη του ευρώ που έχουν απορρόφηση μονάχα 21%. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο θέμα που εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε από την πλευρά της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Δεν είναι δυνατόν να παραμένουν τέτοιες διαφορές απορρόφησης. Θα πρέπει να καταλάβουμε γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές τη στιγμή που είμαστε στον έκτο χρόνο προγραμματισμού το 2012. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι η εξή. <coughs> Αν δούμε αυτά τα στοιχεία βλέπουμε ότι αυτά είναι μονάχα συνολικά στοιχεία. Γιατί υπάρχουν δύο υποπρογράμματα. Υπάρχουν τα λεγόμενα ήπια προγράμματα όταν πρόκειται για την ε, κατάρτιση και τους βοηθάει να βγουν από την ανεργία. Αυτά είναι ήπια προγράμματα. Δεν χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις. Δεν υπάρχει ανάγκη ιδιαίτερης υποδομής αλλά υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο λέγεται υποδομέ. για τους ανθρώπινους σπόρους και βλέπουμε εκεί ότι είναι ακόμα χαμηλότερη η απορρόφηση. 60% εντάξει εν γέννη, αλλά όταν λέμε τι γίνεται για την απορρόφηση στον τομέα αυτό που θέλει κανείς να φτιάξει ένα σχολείο, ένα Ινστιτούτο, πέντε φορές χαμηλότερη είναι η απορρόφηση. Και αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Είναι ο καλύτερος τρόπος τώρα να δίνουμε χρήματα και να επιδοτούμε αυτές τις ενέργειες. Λέμε ότι εκπαιδεύουμε τα άτομα για να έχουν μια θέση εργασία. Μετά από ένα εξάμεινο βγαίνουν από την ε, μαθητεία και την εκπαίδευση, αλλά αν δεν έχουν δουλειά, τι θα κάνουμε, θα του καναβάλουμε μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Αυτό είναι το, <clears throat> το ερώτημα προ την Κομισιόν, γιατί μα δίνεται μονάχα τα συνολικά στοιχεία και τα πράγματα πάνε καλά. Γιατί για αν δούμε τι γίνεται σε σχέση με το Ταμείο Συνοχής και το Περιφερειακό Ταμείο, είναι μόνο 2% καλύτερη η απορρόφηση στο Κοινωνικό Ταμείο. Ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα το που αποκομίζουμε. Πρέπει να σκεφτούμε όμως ποια είναι η ανεργία στην Ευρώπη. Άμα πάνε τόσο καλά τα πράγματα με το κοινωνικό ταμείο. Αλλά δεν μειώνεται η ανεργία παρά το γεγονό ότι πάνε καλά τα πράγματα στο κοινωνικό ταμείο. Επομένως όλη αυτή η ανάλυση δεν έχει νόημα. Εγώ δεν έχω δει λοιπόν τα τελευταία χρόνια που είμαι βουλευτής, τα τελευταία δυόμιση χρόνια ας πούμε, στοιχεία τα οποία να συσχετίζουν την απορρόφηση, την ανεργία και τη δημιουργία θέσεων, νέων θέσεων απασχόλησης. Αλλιώς έχουμε η απορρόφηση 20% που είναι πολλά λεφτά. Είναι μέσα σε 7 χρόνια 50-60 δισεκατομμύρια. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχόμαστε να υπάρχει μια τέτοια έλλειψη σχετισμού. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν μπορώ, θα ήθελα να σταθώ μονάχα στα ουσιώδη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σούριαν και τον κύριο Κοτμάνης για τις ε, συνεισφορές τους. Θα ήθελα να προχωρήσω <clears throat> και λίγο περισσότερο, όπως είπα, και πέρα από τα τρία αυτά άρθρα που έχουν να κάνουν με την ε, εφαρμογή και την απορρόφηση των ε, πόρων. Εγώ κατάλαβα αυτά που ελέγχθηκαν για τα ποσοστά απορρόφησης και ενδεχομένως άλλους δείκτες αποτελεσματικότητας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα πρέπει να δούμε όμως πώς θα αντιδράσουν στη συνέχεια οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Απασχόλησης και αν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια κοινή προσέγγιση <clears throat> με τον εισηγητή από την Επιτροπή ε, Απασχόλησης. Κύριε Σούριαν, εσείς ανησυχείτε για την αύξηση του διοικητικού κόστους. Και εδώ τα πράγματα όμως βαίνουν καλύτερα. Γιατί στο μέλλον θα έχουμε το νέο δημοσιονομικό κανονισμό που ελπίζω θα έχει εγκριθεί πλήρως μέχρι τώρα που θα προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα καταλογίσετε το διοικητικό κόστος και υπάρχουν ήδη μεγαλύτερες προσπάθειες μαζί με την Κομισιόν και το Συμβούλιο για να μην αυξάνει το διοικητικό κόστος και σε ό,τι αφορά την καταποκοπή χρηματοδότηση, αυτό θα συμβάλλει στην μείωση του διοικητικού κόστους ή τουλάχιστον στη μία αύξηση. Εμείς σίγουρα δεν θέλουμε να ε, έχουμε πολλούς οι οποίοι λένε ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκο να υποφεληθούν από τα κονδύλια του κοινωνικού ταμείου, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε μια απλοποίηση του συστήματος, αλλά είμαστε υπεύθυνοι και για να εξετάσουμε το πώς μπορούμε να αποτρέψουμε μια αύξηση της γραφειοκρατίας. Βέβαια, ένα μέρο τη γραφειοκρατία οφείλεται στο γεγονό ότι η διοικητική λειτουργία και παράδοση ακόμα των εθνικών κρατών έναντι τη ε, διοικητική λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ διαφορετικέ. Επομένω, πρέπει κανεί να κάνει διπλή δουλειά. Όταν υπάρχει επιμερισμένη διαχείριση, είναι υποχρεωμένο κανεί να εκπληρεί δύο είδη προποθέσεων και κανόνων. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι γι' αυτό, ώστε τελικά ο τελικός αποδέκτης να μην βρίσκεται σε ένα κικαιώνα εγγράφων, ένα χαρτοβασίλειο που δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει και επομένως αποτρέπεται να προχωρήσει και να εκμεταλλευτεί αυτά τα, αυτά τα προγράμματα και επίσης τον αποτρέπει το γεγονός ότι βλέπει ότι το διοικητικό κόστος αυτής της διαδικασίας και το βάρος το οποίο πρέπει να επομιστεί όλο και αυξάνεται. Εμείς ως Ευρωπαίοι Κοινοβουλευτικοί θέλουμε, <coughs> θα πρέπει να πούμε, ότι είναι δικό μας θέμα να εξασφαλίσουμε ότι θα μειωθεί το διοικητικό άχθος στις επιμερισμένες διαδικασίες διαχείρισης και όχι να αυξηθεί. Γιατί η εμπειρία μας είναι ότι πάρα πολλές φορές αυξάνει, όσο πιο επιμερισμένη είναι μια διαδικασία, αυξάνει πάντα το διοικητικό κόστος. Ο κ. Κοσλόφσκι θέλει μια παρατήρηση να κάνει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ συχνά λέγεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην ουσία είναι μια σωστή πηγή ε, ενίσχυσης αυτών οι οποίοι έχουν ήδη καταρτιστεί, είχαν τη δυνατότητα να έχουν ήδη καταρτιστεί. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις δυνατότητες του ταμείου αυτού με άλλα ταμεία, όπως το FSR, έτσι ώστε τα προγράμματα αυτά να καλύψουν μια ευρύτερη βάση ενδιαφερομένων και να χρησιμοποιούν γι' αυτό πιο συγκεκριμένους δείκτες και κριτήρια στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Επρόκειται για μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων μετά από κάποιες προσανατολιστικές παρατηρήσεις του εισηγητή μας του κ. Γκάιερ δεν θα έχουμε στη διάθεσή μας το κείμενο παρά αργότερα. Έχουμε προχωρήσει θα έλεγα αρκετά γρήγορα. Την 10η Μαΐου θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης του εισηγητή μας. Η προθεσμία είναι η 16η Μαΐου για την κατάθεση των τροπολογιών θα ψηφίσουμε την έκθεσή του στη συνεδρίαση της 19ης και 20ης Ιουνίου, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη για την Επιτροπή Απασχόλησης, η οποία θα ψηφίσει στις 10 Ιουλίου και μόνο τον Σεπτέμβριο η έκθεση αυτή θα φτάσει για ψηφοφορία, συζήτηση και ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Όπως το έχουμε ήδη πει και μετά από αίτημα του εισηγητή θα περάσουμε τώρα στο σημείο 14. Θα μείνουμε πάντα στο κοινωνικό χώρο, αλλά μιλάμε για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ε, η κυρία Ματέρα θα μας παρουσιάσει το θέμα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Ματέρα είναι το πρώτο αίτημα του 12 για την χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και προέρχεται από την Ισπανία. Είναι αίτημα το οποίο κατατέθηκε το 2011, ανταποκρίνεται θα έλεγα ε, στο κλίμα και στη συγκυρία της ε, οικονομικής κρίσης. Μιλάμε για 140 εκατομμύρια ευρώ έτσι ώστε να μπορέσουν να επανακάμψουν στην αγορά εργασίας 1.138 εργαζόμενοι που απολύθηκαν από τον τομέα των κατασκευών ε, στην περιοχή της Βαλένθια. Οι επιχειρήσεις οι οικοδομικές εκεί μείωσαν τις δυνατότητες δανειοδότησης των επιχειρήσεων και των ιδιωτών από πλευράς των τραπεζών, κάτι το οποίο οδήγησε στην πτώση ε, της οικοδομής γενικότερα. Όπως φάνηκε ήδη από το 2011, το Συμβούλιο, παρά τη δική μας ευνοϊκή ψήφο, μπλόκαρε ουσιαστικά τις εξαιρέσει για την χρήση αυτού του ταμείου λόγω ακριβώς της οικονομικής κρίσης. Το ταμείο αυτό κατά κάποιο τρόπο αποκρίνεται μόνο για άμεσες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης όπως μετακινήσεις επιχειρήσεων σε περιπτώσεις συγχρηματοδότησης περιφερειακής κατά 50%. Γι' αυτό και εγώ και έχω εισάγει μια νέα παράγραφο στην έκθεση αυτή. Υπογραμμίζω την ανάγκη που υπάρχει να θέσουμε εκ νέου επιτάπητος με το Συμβούλιο την σημασία να υπάρξει μια επιπλέον παρέκκληση λόγω της οικονομικής κρίσης γιατί μου φαίνεται, αν δεν έχω καταλάβει σωστά αυτά που διάβασα, ότι η οικονομική κρίση δεν έχει βέβαια τελειώσει. Πόσο μάλλον. Σχετικά τώρα με το χρονοδιάγραμμα, 13η Μαρτίου είναι η, κατάθ... η η προθεσμια για την κατάθεση των τροπολογιών, 21η Μαρτίου η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και 28 Μαρτίου η ψηφοφορία στην Ολομέλεια, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γοθμάνης. Υπάρχει κάτι το οποίο για μένα δεν ακόμα σαφής. Μέχρι τώρα το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αντιμετώπιζε περιπτώσεις που χάνει κανείς ανταγωνιστικότητα λόγω της της παγκοσμιοποίησης. Ότι κάποιος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο ανταγωνιστικός, παραδείγματο χάρη. Σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Εδώ, με συγχωρείτε, με το συμπάθειο δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εάν χτίζεται σπίτια και κανείς δεν τα αγοράζει μετά, αυτό δεν έχει να κάνει με την παγκοσμιοποίηση. Είναι απλώς λαθασμένη πολιτική της κυβέρνησης. Δεν είναι σωστό λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σε αυτή την περίπτωση. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσαν τα άτομα τα οποία εργάζονται σε μία επιχείρηση επειδή είναι φθηνότερη η δραστηριότητα αυτή στην Ινδία ή στην Κίνα, αυτό το καταλαβαίνω, ότι έχει να κάνει με την παγκοσμιοποίηση. Αν εσείς χρόνο με το χρόνο κάνετε μια φούσκα στον οικοδομικό τομέα και πιστεύουν οι εργολάβοι ότι κάποιος θα έρθει να, να ζήσει σε αυτά τα σπίτια και στην Ισπανία ακόμα και στους μετανάστες ζητήσαν να μείνουν εκεί πέρα. Εγώ ποτέ δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο λοιπόν. Αυτό είναι λάθος. Ναι, ναι, καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Η κυρία Ανδρέασεν. Και εγώ θέλω να υποστηρίξω αυτά που είπε ο κύριος Γκοντμάνης. Το πρόβλημα στην Ισπανία ήταν ακριβώς ο χώρος της κατασκευαστικής και οικονομικής ε, δραστηριότητας και έχουμε άτομα τα οποία αυτή τη δουλειά μόνο ξέρουν να κάνουν. Πώς θα τους ε, καταρτήσουμε εκ νέου, πώς θα τους μετατρέψουμε. Έχει γίνει μια δραστηριότητα στον οικονομικό τομέα που ήταν στα όρια της νομιμότητας, αν ήταν νόμιμη. Να μετοναθύνουμε λοιπόν κονδύλια για τέτοιες ενέργειες, αυτό είναι λαθασμένο θα οξύνει το πρόβλημα ακόμα περισσότερο. Αυτά τα άτομα δεν έχουν που να δουλέψουν πια, γιατί όλα αυτά τα πράγματα στον οικοδομικό τομέα έχουν τελματώσει, έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Είναι δουλειά της κυβέρνησης, όχι δικιά μας. θα θέλατε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω στον συνάδελφο να πω ότι το αίτημα αυτό ανταποκρίνεται στις παρεκκλήσεις, εξαιρέσεις οι οποίες έχουν γίνει δεκτές στα πλαίσια του κανονισμού του συγκεκριμένου ταμείου από το 2009 λόγω της οικονομικής κρίσης και μιας και η περιοχή της ε, Βαλένσια ζήτησε την κινητοποίηση του Ταμείου όχι για λόγους παγκοσμιοποίησης, αναφέρθηκε στην απώλεια ανταγωνιστικότητας, αλλά αναφέρεται συγκεκριμένα το αίτημα αυτό στα προβλήματα που δημιούργησε η οικονομική κρίση. Ως εκ τούτου ανταποκρίνεται πλήρως στις προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες του συγκεκριμένου ταμείου. Και από τον Ιανουάριο το 2012 θυμίζω ότι όλα τα αιτήματα τα οποία θα γίνουν δεκτά πρέπει να αφορούν εκ νέου αποκλειστικά την παγκοσμιοποίηση, όχι όμως αυτά που κατατέθηκαν στην προηγούμενη περίοδο. Όπως είπε η κυρία Άντρεσεν, ο τομέας της οικοδομής στην Ισπανία είναι σε σοβαρή κρίση. Και πράγματι θα πρέπει η κεντρική κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες ε, απαντήσεις ε, στο πρόβλημα, αλλά το θέμα είναι να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα κοινοτικά μέσα, τα ευρωπαϊκά μέσα. Είναι ένα μέσο το οποίο απευθύνεται στους πολίτες αποκλειστικά. Δεν απευθύνεται στην επανικοδόμηση ας πούμε, επιχειρήσεων ή βιομηχανιών. Και θυμίζω ότι κατετέθη εγκαίρως μετά από τις ψηφοφορίες και τις αποφάσεις τις οποίες ε, εμείς πήραμε. Γι' αυτό παρακαλώ να αλλάξετε την άποψή σας έγκαιρα. Η Γιούτε. Θέλω να υποστηρίξω την Μπάρμπαρα. Ξέρω ότι κάποιοι δεν ενοχλούνται από όλα αυτά. Εμένα με ενοχλούν όλα αυτά και ιδίως επειδή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κρίσης. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να είμαστε όλοι έτοιμοι να βοηθήσουμε τους εργαζομένους όσο βρεθήκαμε έτοιμοι στο παρελθόν να βοηθήσουμε τις τράπεζες στο παρελθόν στις οποίες δώσαμε πάρα πολλά εκατομμύρια. <clears throat> Πρέπει φυσικά οι κανόνες να τηρούνται και <clears throat> αν η Κομισιόν μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι οι κανόνες έχουν τηρηθεί, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε <clears throat> τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν φταίνε αυτοί για την φούσκα ε, στο οικοδομικό τομέα στην Ισπανία. Γι' αυτό υποστηρίζω την πρόταση της Μπαρμπάρα. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βέρτμαν έχει δει στο λόγο, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την Ισπανία, <clears throat> θέλω να πω ότι προφανώς πρέπει να υποστηρίξουμε τους πολίτες στην Ισπανία. Αλλά για την Ισπανία θέλω να κάνω ακόμα μία, παρουσί, ε, μία παρατήρηση για το πού χτιστήκανε αυτά τα κτίρια. Γιατί ορισμένε φορές πολλά από αυτά τα κτίρια ήταν αυθαίρετα, ήταν παράνομα βάση του ισπανικού δικαίου σε σχέση με, την, με το κτίσιμο των σπιτιών σε, στην παραλία, σε, παραθα, σε περιοχές κοντά στη θάλασσα. Οπότε είμαι υποχρεωμένο να υποστηρίξω αυτά τα οποία λέει ο κ. Γκοτμάνης. Θα πρέπει να κάνουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ μιας κρίσης, μιας οικονομικής κρίσης και των αποτελεσμάτων της παγκοσμιοποίησης. Και στην Ισπανία νομίζω ότι είναι σαφή τα πράγματα. Πολύ ωραία. Ναι, θα πρέπει να έχουμε, όπως ε, πει η συγγήτρια, να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια από την 1η Ιανουαρίου 2012. <clears throat> Αλλάζουν και οι κανόνες. Σας υπενθυμίζω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Για να δω, εδώ το είχα, εδώ το είχα λοιπόν. 13 Μαρτίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Η Κομισιόν θα γνωμοδοτήσει στις 14 και στην επόμενη συνεδρίασή μας 21 Μαρτίου της ησημερίας θα ψηφίσουμε. Επομένως θα δούμε τότε τι θα πούν και οι μεν αλλά και οι δε. Ευχαριστώ την εισηγεσία και τώρα περνάμε στο 7 δηλαδή το θέμα για τη διαπραγμάτευση του, δημοσιο... του δημοσιονομικού παλαισίου. Καταρχήν να δούμε τι είπε η ομάδα επαφής την περασμένη εβδομάδα και μετά θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, όπως γνωρίζετε λέγω το Κοινοβούλιο συνέστησε μια αρκετά ιδιαίτερη διαδικασία για να παρακολουθήσει αυτή τη διαπραγμάτευση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και για να διασφαλίσει έτσι το συντονισμό με την εργασία και των υπολείπων κοινοβουλευτικών επιτροπών που χρειάζεται να εξετάσουν και να προετοιμάσουν την ψηφοφορία όλων των νομοθετικών κειμένων που βασίζονται στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων που προβλέπει αυτό το πολιετές ε, πλαίσιο. Υπό την Προεδρία του κυρίου Σούλτς, Προέδρου του Κοινοβουλίου και αποτελείται από τα μόνιμα μέλη που είναι η ομάδα της Κομπούς που διαπραγματεύεται το πολιετές πλαίσιο και από την άλλη οι συντονιστές και συντονίστριές μας ώστε όλες οι πολιτικές ομάδες να συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση αυτή. Εκτός αυτών, ανάλογα με τις συνεδριάσεις καλούνται και άλλοι βουλευτές, ίσως και εκπρόσωποι της Κομισιόν, εφόσον η διαπραγμάτευση το απαιτεί και καθώς θα προχωράει. Κατά την τελευταία συνεδρίασή τους, ο πρόεδρος Σούλτς κάλεσε τους προέδρους των κυριωτέρων κοινοβουλευτικών επιτροπών που δαπανούν κονδύλια και που ενδιαφέρονται από τον πολιτισμό, δηλαδή γεωργία, αλληλεία, ήτρε, περίφ, μεταφορές και απασχόληση. Άλλοι δε πρόεδροι θα προσκληθούν εν καιρό το δέοντι και εν ευθέτω χρόνο. Ένα από τα θέματα που εξετάστηκαν ήταν και το κατά πόσον ή μάλλον το πώς θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις αυτές παράλληλα με όλες αυτές τις επιτροπές που δαπανούν χρήματα. Δηλαδή το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων απαιτούσε ή όχι παράλληλη διαπραγμάτευση. Μήπως το νομοθετικό στοιχείο προέχει η συνένεση στην οποία καταλήξαμε τελικά ήταν να ενθαρρύνουμε την νομοθετική δουλειά καλώντας τις επιτροπές να μην βάλουν αριθμούς ακόμη διότι αν κάθε επιτροπή έβαζε από τώρα αριθμούς για τον προϋπολογισμό που θέλει να δοθεί στην ΚΑΠ, στην περιφερειακή πολιτική κτλ. Αν άρχιζαν από τώρα λέγω με τους αριθμούς τότε θα χανόταν κάθε ενδιαφέρον για συντονισμένη διαπραγμάτευση και κάθε επιτροπή θα είχε τον πειρασμό να παίρνει άτεγκτη και μαξιμαλιστική θέση με τον κίνδυνο επομένως έτσι να υπονομευτεί η συνολική θέση του Κοινοβουλίου στον προϋπο, στην διαπραγματεύση του προϋπολογισμού. Γι' αυτό οι επιτροπές πρέπει όσο μπορούν περισσότερο να διαπραγματευτούν τα πράγματα ως προς το νομοθετικό περιεχόμενο, το πολιτικό περιεχόμενο της ΚΑΠ ας πούμε ή τον κανονισμό για το κοινωνικό ταμείο για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως κλπ. Αλλά αλλά να περιμείνουν πριν βάλουμε και εμείς αριθμούς. Ο πρόεδρος Σούλτς προτίθεται να έρθει την επόμενη εβδομάδα για να μιλήσει για αυτό το βασικό θέμα με το σύνολο των Προέδρων των Επιτροπών στην επόμενη διάσκεψή των στο Στρασβούργο, όπως γίνεται κάθε Τρίτη Στρασβούργο. Οι συγητές λοιπόν των διαφόρων επιτροπών βρίσκονται συνεχώς σε επαφή μεταξύ τους, έχουν συνεννοηθεί ήδη, έχουν αρχίσει να συνεννοούνται και ο πρόεδρος Σούλτς μας ανακοίνωσε ότι προτίθεται επίσης με κάθε ευκαιρία να, συναντιέται, να συναντηθεί με το Συμβούλιο, την Προεδρία ή τα μέλη του, για να του υπενθυμίσει τις κυριότερες θέσεις και απαιτήσει και αιτήματα του Κοινοβουλίου. Ήδη στο Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας το έπραξε και μας έστειλε το κείμενο της παρέμβασης του εκεί υπάρχει, δεν ξέρω αν έχει διανεμηθεί σε όλους, εκεί ιδίως αναφέρεται μία παράγραφος ειδικά για τον προϋπολογισμό. Μίλησε πολύ γενικά, αυτό είναι φυσικό σε αυτή τη φάση, γιατί η διαπραγμάτευση για το πολιετές πλαίσιο δεν ήταν το θέμα του Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας. Αντίθετα, θα είναι ένα από τα κυριότερα θέματα του τον Ιούνιο και αυτή τη στιγμή προετοιμαζόμαστε για την επόμενη και σημαντικότερη αυτή φάση του, των εργασιών του Συμβουλίου τον Ιούνιο. Μέχρι τότε και ανάλογα με τις συναντήσεις που θα γίνουν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο με το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα δούμε οι συγητές θα μας προτείνουν θα μας δούνε αν πρέπει, αν χρειάζεται και αν είναι πότε να ενημερωθούμε ή να τροποποιήσουμε την εντολή, τη διαπραγματευτική εντολή που μας έδωσε η Ολομέλεια για την έκθεση ΣΟΥΡ και αν χρειαστεί αυτό θα το πράξαμε στα πλαίσια ενός νέου ψηφίσματος που θα επεξεργαστεί η Επιτροπή Προϋπολογισμών στην και θα προτείνει στην Ολομέλεια τον Μάιο ή τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να το δούμε. Βασικά όμως αυτό αποφασίστηκε. Τέλος, Μιλήσαμε και για την προετοιμασία της διάσκεψης για το πολιετές αυτό πλαίσιο διαθεσμικής αλλά και διακοινοβουλευτικής διάσκεψης που θα γίνει στις 22 Μαρτίου σε 15 μέρες περίπου δηλαδή και που θα είναι η δεύτερη του είδους της. Θα θυμάστε ίσως ότι με δική μας πρωτοβουλία και σε συμφωνία με την Πολωνική τότε Προεδρία έγινε μια πρώτη τέτοια διάσκεψη τον περασμένο Οκτώβριο. Αυτή τη φορά, λίγους μήνες αργότερα, οι διαπραγματεύσεις ή ανταλλαγές απόψεων, γιατί δεν άρχισε ακόμα η διαπραγματεύση, οι ανταλλαγές απόψεων πολλαπλασιάστηκαν και αρχίζουν και να εμβαθύνονται και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτή τη στιγμή να τις διευρύνουμε στο και στους εθνικούς βουλευτάς και θα καλέσουμε γι' αυτό τους εκπροσώπους των 27 και των 27 κυβερνήσεων άρα η διαδικασία της διαπραγμάτευσης που αρχίζει τώρα η δική μας αντιπροσωπεία θα συναντήσει και την Τρόικα των Προεδριών και στις 22 Μαρτίου εκπροσώπους των 27 κυβερνήσεων. Θα συναντήσουμε δηλαδή και εκπροσώπους κυβερνήσεων και εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στις Εθνικές Βουλές για να εκφράσουν και αυτή την άποψή τους για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τις προτεραιότητές του και να δούμε τι φρονούν για τη χρηματοδότησή του. Θέλουν να διατηρηθεί το υπάρχον σύστημα, θέλουν να αλλάξει, να υπάρξουν νέοι ήδη πόροι. Αν η πρόταση της Κομισιόν για τους νέους αυτούς ιδίους πόρους ε, τους βρίσκει σύμφωνους ή αν υπάρχουν διαφωνίες. Όλα αυτά θα τα δούμε στη διάσκεψη αυτή της 22ης Μαρτίου. και θα δούμε με τι ερωτηματολόγιο, με τι, ποια θα είναι ακριβώς μάλλον η ημερήσια διάταξη. Αυτά για τα σεπαφάς. Ε, προτείνω τώρα στον Ράιμερ Μπέγκε αν θέλει να προσθέσει τίποτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχω να προσθέσω ουσιαστικά τίποτα γιατί παρουσίασε τα πορίσματα της ομάδος επαφής ο πρόεδρος μας Νομίζω ότι είναι θετικά αυτά τα πορίσματα <clears throat> και είναι πολύ καλός τρόπος να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και να έχουμε μια μορφή συντονισμού <clears throat> για τα θέματα του προϋπολογισμού. Θέλω να προσθέσω ότι ο εισηγητής ε, για τις δημοσιονομικές προοπτικές της επόμενης περίοδου κάθε πέμπτη πρωί θα είναι σε επαφή με την ομάδα επαφής και θα έχει τακτικές ανα, ανταλλαγές απόψεων όσοι θέλουν λοιπόν ε, να ασχοληθούν ε, με αυτά τα θέματα πρέπει να ξέρουν ότι ο εισηγητής προσκαλείται όταν αυτό είναι απαραίτητο από την ομάδα επαφής. Επίσης ο Αλάν μας είπε ότι η ομάδα επαφής είχε ήδη επιτύχει μία συνένεση σε αυτό το χρονικό επίπεδο να μην αναφέρει καθόλου αριθμητικά στοιχεία για τα κονδύλια στα πλαίσια των επομένων δημοσιονομικών προοπτικών. Εγώ νομίζω ότι αυτός είναι και ο σωστός δρόμος. Ξέρω ότι κάποιοι έχουν ε, διαφορετικές εκτιμήσεις για αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να συζητηθεί το θέμα αυτό και από τη συνέλευση των Προέδρων και των πρόεδρων των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ώστε με τον τρόπο αυτό να μπορούμε να έχουμε μια ενιαία γραμμή χωρίς διαμάχες μεταξύ μας. Νομίζω ότι και ο κύριος Κάλφιν είχε την ίδια αντιμετώπιση. Εμείς ως εισηγητές δεν είχαμε καθόλου πρόβλημα να δώσουμε στοιχεία για τα 72 προγράμματα τα οποία βρίσκονται στην ε, συναπόφαση. Αλλά πού θα μας πήγαινε κάτι τέτοιο. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαμάχες. Γι' αυτό Πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουμε στην ε, πιο σόφρονα γραμμή η οποία δεν θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα και να αφήσουμε αυτή τη διατύπωση που υπάρχει. Ένα δεύτερο στοιχείο που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο είναι και πρέπει να είναι σαφές αυτό σε όλους ότι συμφωνούμε όλοι ότι η προετοιμασία των νομοθετικών ε, ε δραστηριοτήτων και νομίζω ότι στα πλαίσια αυτά δεν χρειαζόμαστε την προηγούμενη ε, συμφωνία διαθεσμικού χαρακτήρα. Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει η πρώτη ανάγνωση στην Ολομέλεια χωρίς ενδεχομένως να ληφθεί μια απόφαση γιατί αν καταλήξουμε σε διαφορετικές ε, διαδικασίες <clears throat> κάποιες θα προχωρήσουν πιο γρήγορα γιατί είναι οι λιγότερο πεπλεγμένες αν καταλήξουμε σε μερικές και αποσπασματικές συμφωνίες, δεν θα μπορούμε να έχουμε συνοχή σε αυτά που κάνουμε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια ενιαία γραμμή. Δεν μπορεί η γραμματεία μας να τα σχεδιάσει όλα και να τα έχει όλα στο μυαλό της. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και οι ψηφοφορίες στην Ολομέλεια θα πρέπει να έχουν κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τον Ιούνιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο, οτιδήποτε τέτοιο. Και επίσης ήρθα σε επαφή με ένα εκπρόσωπο της Δανικής Προεδρίας, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εκεί πρέπει να επιμείνω σε δύο σημεία. Και αυτό και έναντι της Κομισιόν, με τους οποίους έχουμε μιλήσει, ώστε δεν πρέπει να έχουμε μονάχα πρόσβαση στα δημοσιονομικά δελτία που μας δίνουν για ορισμένα προγράμματα, αλλά να έχουμε μια πληρέστερη πληροφόρηση για το τι υπάρχει πίσω από αυτά τα προγράμματα. Γιατί η ομάδα αυτή των φίλων της Προεδρίας συζητά για όλα αυτά τα θέματα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη συζήτηση. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γνωρίζουμε τι συζητάτε και να έχουμε και μια καλύτερη ιδέα και για τα αριθμητικά ποσά τα οποία αναφέρονται. Αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο σε πολιτικό επίπεδο και πρέπει να το πούμε σαφώ στην Κομισιόν. Γιατί θα πρέπει να βρισκόμαστε σε επίπεδο ισοτιμίας και με το Συμβούλιο. Και επίσης, και αυτό έχει γίνει δεκτό, να γνωρίζουμε και τις θέσεις της Προεδρίας σε σχέση με τη διαπραγμάτευση με το Κοινοβούλιο για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων αναφέρει ένα λεγόμενο κοιτία διαπραγματεύσεων, αλλά αυτό δεν μας δίνει αρκετή πληροφορία για να ξέρουμε τι ακριβώς προβλέπεται. Μας ενδιαφέρει να ξέρουμε ποιες είναι οι συζητήσεις στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, ώστε να έχουμε και εμείς μια εμπεριστατωμένη ε, θέση για αυτά τα θέματα. Έτσι θα αποτρέψουμε τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο να ανακύψει ένα πρόβλημα και να καθυστερήσει η διαδικασία για την έγκριση των δημοσιονομικών προοπτικών. Θέλω λοιπόν και πάλι να κάνω μια έκκληση στη Δανική Προεδρία να μας αναφέρει τις σκέψεις της εγκαίρως ώστε να μπορέσει να τα επεξεργαστεί με τον κατάλληλο τρόπο και η ομάδα επαφής και η Επιτροπή Προϋπολογισμών και όχι μόνο την τελευταία στιγμή να γνωρίσουμε περί τίνος πρόκειται, γιατί αυτό θα μας οδηγήσει σε δυσκολίες. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ, Ράιμερ. Νομίζω ότι ξεκαθάρισε τα πράγματα. Ο Ζαν Λουκ θα ήθελε κάτι να συμπληρώσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά που μπορεί να προσθέσει κανείς. Υπάρχει το σχέδιο γνωμοδότησης που έχει ήδη προταθεί και που θα συζητήσετε. Εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τη συνεδρίαση της 22 του μηνός, γιατί φοβάμαι ότι μέχρι τότε δεν θα έχουμε το έγγραφο που έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μας δίνει μια πλήρη εικόνα. Δηλαδή τι σημαίνει μείωση της συνεισφοράς επί τη βάση του εθνικού ακαθάριστου. Και εφόσον δεν έχουμε το έγγραφο αυτό, η συζήτηση με τα κοινοβούλια των κρατών μελών είναι μια δύσκολη συζήτηση, η οποία μπορεί να στρίψει άσχημα προς ιδεολογικά επίπεδα και να μην είναι μια τεκμηριωμένη πραγματιστική συζήτηση. Θα ήθελα να σημειώσω ότι Είχα πρόσφατα μία συνάντηση με τον εκπρόσωπο της Δανικής Προεδρίας που προεδρεύει της Ομάδας Εργασίας για τους Ιδίους Πόρους και μου είπε ότι στα πλαίσια του πακέτου για τον Ιούνιο θα συμπεριλάβουν τους ίδιους πόρους, έτσι ώστε να μην αντιμετωπιστούν με ξεχωριστό τρόπο. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο μπροστά μας, αλλά η Προεδρία συνδέει τα θέματα αυτά και δεν θα έχουμε τον κίνδυνο να συζητάμε μόνο τις δαπάνες στη συνάντηση κορυφής του Ιουνίου, αποφεύγοντας αν θέλετε και κάποιες πολύ ριζικές σε βάθος συζητήσεις αποκλειστικά για τους ίδιους πόρους. Ευχαριστώ Ζων Λουκ. Συμπληρώνοντας αυτά τα οποία είπε ο Ζων Λουκ σχετικά με τους αριθμούς εισαγωγικά, που ζητά ο Ζαν Λουκ Ντοάν από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και μήνες. Ποιες θα είναι δηλαδή οι συνέπειες για κάθε ένα από τα κράτη-μέλη της μείωσης των εθνικών συνεισφορών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για νέες προτάσεις στο τομέα των ιδίων πόρων. Αυτό θα ακουγόταν ενδιαφέρον για τα κρατη και, ε, και τα κοινοβουλιά τους. Μετά από συζήτηση με τους συντονιστές έστειλα μία επιστολή στον Λεβαντόφσκι, τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι, για να είναι παρόν στη συνάντησή μας στις 21 Μαρτίου, ε, την παραμονή δηλαδή της συνάντηση στις 22 Μαρτίου. Θα έρθει λοιπόν εδώ για μία και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση και στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής θα μας δώσει αυτούς τους αριθμούς και θα μας μεταφέρει και όλα τα αριθμητικά στοιχεία που έχει σχετικά με την κατανάλωση την απορρόφηση των πιστώσεων πληρωμών για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε σωστά τις διαπραγματεύσεις για το 2013 για τις πιστώσεις πληρωμών και του διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2012, γιατί από ό,τι φαίνεται η κρίση στις πιστώσεις πληρωμών ήδη από φέτος θα πάρει διαστάσεις πολύ μεγάλες. Θα έχουμε λοιπόν τα στοιχεία αυτά την παραμονή της 22ης Μαρτίου. Δεν ξέρω αν θα τα διανύμουμε και στους συμμετέχοντες στις 22 του μηνός θα δούμε αυτά. Τι θα κάνουμε ακριβώς. Να προσθέσω ότι εφόσον ο Ράιμερ συμφωνεί θα προτείνω να προσκληθεί στη συνεδρίαση της διάσκεψης των Πρόεδρων Επιτροπών με τον Ιβάη Λοκάλφιν και άλλους συγητές την επόμενη εβδομάδα γιατί εκεί θα είναι παρόν ο Σούλτς που θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της ομάδας επαφής. Λοιπόν, έχουν ζητήσει και άλλοι το λόγο. Φέρμε. Γιώραν Φέρμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώς ο Ιβάιλο Καλφίν είναι στην Ελλάδα σε μια σημαντική αποστολή, δεν είναι ανάμεσά μας. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του προσωπικά, αλλά μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της ομάδας μου και είχαμε μεγάλες συζητήσεις στην ομάδα μας για τα θέματα αυτά. Συμφωνούμε με τη στάση του Ράιμερ και με αυτά που είπατε, Πρόεδρε. Αυτό που έχει σημασία είναι η μεγάλη πλειοψηφία που έχουμε πίσω από την ε, Επιτροπή ΣΟΥΡΕ που αντιπροσωπεύει το 80% των μελών του σώματος πρέπει να διατηρηθεί. Αν χάσουμε την πλειοψηφία αυτή τότε θα χάσουμε και τις δύο διαπραγματεύσεις. Απαιτείται η πλειοψηφία αυτή και στη διαδικασία συνένεσης. Αν πράγματι είμαστε ισχυροί εκεί με το Συμβούλιο θα το πετύχουμε. Μια βασική απειλή είναι να μην πετύχουμε τη συνένεση, ίσως αν υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία, αλλά από την άλλη το να σπάσουμε τη συζήτηση που θα μπορούσε, κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι καλό για κάποιες πολιτικές ομάδες, για κάποιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Η αποσπασματική αντιμετώπιση δηλαδή δεν είναι η σωστότερη. Εγώ δεν θέλω να πω στις επιτροπές μας και στις πολιτικές μας ομάδες το πώς θα δουλέψουμε αλλά παρόλα αυτά διατρέφουμε τον κίνδυνο το Συμβούλιο να επιλέξει συζήτηση σε τομείς που είναι ζωτικοί για αυτούς και να αγνοήσει άλλους τομείς οι οποίοι είναι ζωτικοί για μας. Λοιπόν, απαιτείται εδώ ε, πειθαρχία και απαιτείται να μην υποκύψουμε στις τομεακές προτάσεις, στις αποσπασματικές προτάσεις του Συμβουλίου γιατί θα σπάσουν την πλειοψηφία που έχουμε στο σώμα. Εγώ είμαι υπέρ της περαιτέρω ανάλυσης των αριθμητικών στοιχείων που ανέφερε και ο Ζαν Μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω αναλύσεις για το τι σημαίνει η έκθεση Σούρε. Μπορούμε να κάνουμε βήματα προόδου και εκεί ε, στην πιθανή ανάλυση σαν παράδειγμα του τι θα σημαίνει η μη επίτευξη της συνένεσης κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε το Κοινοβούλιο επί τη βάση αριθματικών στοιχείων γιατί αυτό θα ήταν καταστροφικό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση και σε επίπεδο διασκέψεως Προέδρων Πολιτικών Επιτροπών και Προέδρων Πολιτικών Ομάδων αν χάσουμε το σύνολο στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, δεν θα πάνε καλά τα πράγματα, γι' αυτό συμφωνώ με τον Σούλτς και με εσά και θα πρέπει να τεθεί σωστά το θέμα και στη διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών και στις Προέδρους των πολιτικών ομάδων. Για το θέμα αυτό λέω, Πρόεδρος. Ξέχασα να σας πω κάτι το οποίο είναι κεφαλαιόδες, πιστεύω. Ότι το Συμβούλιο βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με εμάς. Προφανώς. Προφανώς. Δηλαδή, οι Υπουργοί Γεωργίας ε, θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν με την Επιτροπή της Γεωργίας για να έχουν το μέγιστο χρηματοδότηση για το δικό του τομέα. Δηλαδή και το Συμβούλιο έχει προβλήματα εσωτερικής οργάνωσης όπως και εμείς και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στο παρελθόν οι διαπραγματεύσεις ξεκινούσαν από μια κοινή δήλωση όλων των θεσμικών οργάνων για να παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία που προ... προηγουμένως περιέγραψα. Και στην ομάδα εργασία εμείς παρουσιάσαμε ένα προσχέδιο κατά κάποιο τρόπο, ένα κείμενο το οποίο θα είναι ενδεικτικό για μια κοινή διαθεσμική δήλωση, ώστε να, εξασφαλίσουμε ότι μόνο στο τέλος θα γίνει η διαπραγμάτευση των συγκεκριμένων αριθμητικών ποσών, αριθμητικών στοιχείων. Η αρχική αντίδραση βέβαια σε αυτή την πρόταση ήταν αρκετά αρνητική, γι' αυτό δεν συνεχίσαμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αφήσαμε το θέμα ανοιχτό, αλλά κατά την άποψή μου αυτό το οποίο θα γίνει στην πραγματικότητα είναι ότι θα μας ζητήσει και σε εμά το Συμβούλιο μια τέτοια δήλωση, γιατί τη χρειάζονται όσο και εμείς. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πάρα πολύ γρήγορα, αν μπορούμε όλε αυτές τις αρχές να τις καταγράψουμε σε κάποιο κείμενο και να προχωρήσουμε σε μία επίσημη δέσμευση ή αν θα συνεχίσουμε σε μία άτυπη διαδικασία. Συνεχίζω με τους εισηγητές. Ο Γκέραν ήταν ένα είδος σκιώδης εισηγητού και δίνω το λόγο στην Άννη. Λέω και εγώ από τη δική μου πολιτική ομάδα ότι υποστηρίζουμε αυτή τη γραμμή να είμαστε ενωμένοι, να βασιστούμε στην έκθεση της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ Και πέραν αυτών που είδαμε την τελευταία φορά που κάναμε τη διαπραγμάτευση των δημοσιονομικών προοπτικών, νομίζω ότι όλοι κατανοούν ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι απλώς ένα σημείο αφετηρίας. Στο Συμβούλιο επίσης υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Αυτοί που θέλουν να περικόψουν, θέλουν να περικόψουν κατά 10%. Στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ είχαμε μια καλή συζήτηση με τους αρμόδιους επιτρόπους, με πολλά άτομα από τις επιμέρους ειδικευμένες επιτροπές στο Κοινοβούλιο, με την σωστή με την πάρα πολύ σωστή ηγεσία της Ιούτα και επομένως μπορούμε να ξέρουμε τι είναι αυτά τα οποία μας προτείνει η Κομισιόν και αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό αντανακλούν αυτά που ήδη είχαμε συζητήσει στην Επιτροπή Σούρε. Δεν είναι λοιπόν ότι αυτά τα οποία θα μας προταθούν απέχουν παρασάγκας από αυτά που είχαν συζητήσει οι αρμόδιες επιτροπές. Έχουμε κάποιους εκπροσώπους από τέτοιες επιτροπές, αλλά θα ήταν πραγματικά παράδοξο να είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τελική απόφαση. την άποψή μου δεν είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσουμε κάποια απόσταση και να πούμε ότι θα συζητήσουμε το περιεχόμενο και τα αντίστοιχα θέματα θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή, αλλά δεν θα κάνουμε την τελική συζήτηση στην Ολομέλεια. Δεν προχωρούμε στις διαπραγματεύσεις, δεν βάζουμε αριθμητικά ποσά. Μέχρι στιγμής τα μόνα αριθμητικά ποσά που αναφέρονται είναι η ενδεικτική στόχη, η ενδεικτική πόρη της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ και αυτά δεν μπορούμε να τα παρακάμψουμε όσο το Συμβούλιο δεν έχει εκφραστεί σε σχέση με τις προτάσεις της Κομισιόν. Γιατί κυκλοφορούν και στο Συμβούλιο διαφορετικές ιδέες. Ίσως δεν είναι μονάχα αυτοί που θέλουν να περικόψουν τις δημοσιονομικές προοπτικές, Μπορεί να υπάρχουν και άλλες απόψεις. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις και στο Συμβούλιο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και ευαίσθητη κατάσταση όπου πρέπει να εμπλακούν πάρα πολλοί φορείς, πάρα πολλά όργανα και πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε δροσεροί και ψύχρεμοι και να κρατήσουμε την προσέγγιση της Επιτροπής Σούρε μέχρι ότου έχουμε νέα φρέσκα στοιχεία. Βεβαίως λέει ο πρόεδρος Λαμασούρ. Να σας κάνω μια στρατιωτική σύγκριση. Βέβαια στρατιωτικά θέματα εδώ σε μια Ευρώπη της ειρήνης και τα λοιπά δεν είναι πια της μόδας, αλλά να. Το κατόρθωμα της Επιτροπής ΣΟΥΡ είναι ότι ακριβώς πέτυχε αυτή την πλειοψηφία του 80%. Πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουμε ενωμένοι όσο δυνατόν περισσότερο. Αν ξαφνικά φύγει ένας μεμονωμένος καβαλάρης θα καταστραφούν όλα. Και μάλιστα θα υποχωρήσουμε ένα τάκτος πριν ακόμη συναντήσουμε τον εχθρό κατά μέτωπον. Έχουμε λοιπόν προφανώς συμφέρον να παραμείνουμε ενωμένοι όσο δυνατόν περισσότερο. Όταν δεν θα αρχίσει η μάχη θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και τότε ίσως να μην είναι πια 80% η πλειοψηφία, αλλά πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Αυτό είναι το δυσκολότερο στην πολιτική υπομονή. Πρέπει πάντως να παραμείνουμε ενωμένοι και βλέπω ότι προς το παρόν υπάρχει μεγάλη συνένεση. Λοιπόν, ο James Ellis. Είναι δύσκολο να έχει κανείς υπομονή όταν είναι και παθιασμένος. Εγώ θα κάνω μία σύγκριση με το πνεύμα της, ε, που αφορά τη συνεννόηση με τους εθνικούς βουλευτάς. Είναι πολύ σημαντικό και αυτοί να είναι μαζί μας και όχι εναντίον μας. Μία Ινδική αρχή είναι, λέει, ότι πρέπει να τους πείσουμε να είναι μαζί μας ακόμη και αν δεν έχουν συνείδηση του γεγονότος αυτού ότι είναι μαζί μας δηλαδή. Εγώ είχα το αίσθημα ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε δυνατότητα για τα εθνικά κοινοβούλια να εκφράσουν και αυτά την άποψή τους και όταν συναντιόμασταν είχαν πολύ αρνητική στάση, αυτό είδα εγώ. Τις προάλλες όμως στο ημικύκλιο με τον Βαρόσο και Βανρομπούι ε, είχαν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή είδαμε ότι υπήρχε η δυνατότητα να εκφραστούν και αυτοί και είχαν ήδη πει ρωτήσει αν στις 22 Μαρτίου θα μπορούν επίσης να εκφραστούν Δεύτερον, κάτι ουσιώδες, ο Μπαρόζο είχε δίκιο. Δηλαδή, μιλάμε πολύ εδώ μέσα για το 2020. Ποτέ όμως δεν άκουσα έναν υπουργό της χώρας μου ή άλλης χώρας να εκφράζεται για αυτό το θέμα. Γίνονται λοιπόν από τη μια μεριά συζητήσει στα ευρωπαϊκά όργανα και από την άλλη στα εθνικά κοινοβούλια και λένε τα ίδια για την ανάπτυξη και την αναπασχόληση αλλά δεν θα μπορούσαμε με την ευκαιρία της 22ης Μαρτίου να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη και ιδίως τους αρχηγούς των κυβερνήσεων αλλά και τους υπουργούς και άλλους βουλευτές να μιλήσουν και αυτά για το πρόγραμμα αυτό του 2020 αυτό το λέω έτσι απλώς για να κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των ε, δημοσίων χρημάτων. Ευχαριστώ, James. Συμφωνώ απόλυτα και με τα δύο. Τώρα, για το πνεύμα της διάσκεψης της 22ης Μαρτίου, πήραμε μαθήματα από την προηγούμενη εμπειρία της 20ης Οκτωβρίου, που ήταν και η πρώτη φορά, και τα κοινοτικά θέματα ήταν κυρίαρχα, ιδίως την πρώτη ημερίδα όπου η Κομισιόν είχε την ιδέα που είναι θεωρητικά ενδιαφέρουσα αλλά που αποδείχτηκε καθόλου πρακτική να δοθεί κυρίως ο λόγος σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλους που ενδιαφέρονται από τον προλογισμό. Αυτό δεν ήταν πολύ ενδιαφέρον και έφαγε το 1 τρίτο του χρόνου της διάσκεψης υπέρ ομιλητών που δεν ήταν εκλεγμένοι, δεν ήταν βουλευτές. Είτε Ευρωπαίοι, είτε Υπουργοί, είτε Εθνικοί βουλευτές. Και αυτή τη φορά το σύνολο του χρόνου θα αφιερωθεί στους βουλευτές. Και στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που θα θελήσουμε να φυγούν δηλαδή. Ελπίζουμε να ακουστούν οι εκπρόσωποι όλων των πολιτικών ομάδων. Για το δεύτερο που είπε ο Τζέιμς, πράγματι και εγώ βλέπω στη χώρα μου και νομίζω το ίδιο θα ισχύει σε πολλές άλλες, ότι η Ευρώπη του 2020 είναι ένα θέμα με το οποίο δεν ασχολείται καμία κυβέρνηση και το κάνουν επίτηδες, δεν θέλουν να ασχοληθούν. Θεωρούν δηλαδή ότι δεν τους αφορά. Αυτό είναι περίεργο, διότι μετά από όλες τις κρίσεις υπερχρέωσης και αφού υπογράφει και η νέα συνθήκη Fiscal Compact, πώς το λένε, τέλο πάντων, και όλοι λένε ότι δεν αρκεί η λιτότητα, χρειάζονται και επενδύσεις, τι κάνουν στην ουσία ξαναλένε αυτά που λέει το πρόγραμμα 2020 με το οποίο δεν θέλουν να ασχοληθούν. Στις 22 Μαρτίου λοιπόν θα το δείξουμε αυτό για να πούμε ότι το ίδιο είναι αυτό που λένε αυτοί και αυτό που λέει το 2020. Έχει δει και ο Τζέιμς που μας, υποστηρεί, που μας υπενθυμίζει ότι τα εθνικά κοινοβούλια και κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται για το 2020. Πρέπει λοιπόν να τους υποδείξουμε ότι είναι ακριβώς αυτό που ζητάνε. Η Χέλγα Τρούπελ. Ευχαριστώ πολύ, αλλά θέλω να αναφερθώ στα απορίσματα της τελευταίας συνάντησης της ομάδας επαφής. Ο πρόεδρος Σούλτς είπε πολύ σαφώς ότι η κοινή μας θέση είναι ότι είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο, αλλά μπορούμε ακόμα και να αντιπαρατεθούμε με το Συμβούλιο, να αγωνιστούμε εναντίον του. Ο στόχος του Κοινοβουλίου είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα περάσουν οι θέσεις <clears throat> της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ, η οποία είχε μια πλειοψηφία 80% που υποστηρίχθηκε. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή μας. Δεν θα, υποστη... Δεν θα υποχωρήσουμε από αυτή. Αν χάσουμε λοιπόν αυτή τη θέση, και δεν μπορέσουμε να κρατήσουμε συντεταγμένες τις λεγεώνες μας, τότε έχουμε χάσει, το, έχουμε χάσει τη μάχη. Και μετά από αυτά που συζητήσαμε με αρχηγούς, με επικεφαλής ε, ε, επιτροπών στην ομάδα επαφής, νομίζω ότι το μπαλάκι έχει έρθει στις πολιτικές ομάδες που είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το δεσμευτικό πλαίσιο είναι αυτό που επετέχθη από την Επιτροπή Σούρε. Κάποιοι συνάδελφοι δεν το έχουν κατανοήσει αυτό απόλυτα. Ψήφισαν αυτή την έκθεση όπως ψηφίσουν πολλές άλλες εκθέσεις. Αλλά κανείς από αυτούς δεν διάβασε την έκθεση και δεν κατάλαβε ποια είναι τα στρατηγικά στοιχεία αυτής της έκθεσης και επομένως ότι είναι απαραίτητο να παραμείνουμε ενωμένοι και να βάλουμε σε δεύτερο <clears throat> επίπεδο τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και συμφέροντα κάθε επιτροπής στο όφελος της διατήρησης τη ενότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια μεγάλη πλειοψηφία που θα υποστηρίξει την κοινή θέση. Και τώρα μπορώ να έρθω στο θέμα του πώ, με το Συμβούλιο και ιδίως με τη συνδιάσκεψη που θα γίνει τώρα το Μάρτιο, πώς θα διαμορφωθεί μια στρατηγική. Υπάρχει αυτή η πρόταση λοιπόν μείωση κατά 10% από τις χώρες οι οποίες είναι καθαροί πληρωτές είπανε άδεια είναι τα ταμεία μας. Δεν μπορούμε στο κράτος μας να πληρώνουμε πώς θα μπορέσουμε να δίνουμε κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε την εντύπωση ότι επιχειρηματολογούμε λόγω εγωιστικού συμφέροντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Ότι είμαστε οι ευρωκράτες που περνάμε πάντα καλύτερα από ό,τι στα κρατη Όλη αυτή η συζήτηση λοιπόν για, τον ε, προϋπολογισμό μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν καταφέρουμε να, δείξουμε ότι είναι προς το συμφέρον όλης της Ευρώπης να μην υπάρξει αυτή η περικοπή κατά 10% στις χώρες που είναι καθαρή συνεισφορής. Οπότε το βασικό ερώτημα των δημοσιογράφων που λέει πώς εσείς υποστηρίζετε τι προτάσει τη Κομισιόν όταν δεν υπάρχουν λεφτά για να, για χρηματοδοτήσουμε τους Ιλλανδούς ή τους ε, Πορτογάλους. Η δική μου απάντηση είναι όταν υπάρχουν κοινοτικά κονδύλια, όταν υπάρχει ευρωπαϊκός Προπολογισμό, έχει ένα πιο θετικό αποτέλεσμα από ότι όταν δεν υπάρχει. Μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το επιχείρημα και να γίνει σαφέ ότι αν υπάρχει υψηλότερος ευρωπαϊκός ε, προπολογισμό έχουμε καλύτερο συνολικό αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύτερη αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, καλύτερες υποδομές για την ενέργεια και την πιο πράσινη οικονομία και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών οικονομικών δραστηριοτήτων. Κανένα από τα κράτη-μέλη μας δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικό, τόσο επιτυχημένο με την πολιτική ανταγωνιστικότητα στα τελευταία χρόνια όπως το θέλαμε. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να επιτύχουμε νέους στόχους και κριτήρια ανταγωνιστικότητας και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω ότι τώρα πρέπει να υπάρξει μια κοινή απόφαση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου να υπάρξει μια κοινή στρατηγική ανταγωνιστικότητας εν ώψη των στόχων της Ευρώπης 2020. Πρέπει λοιπόν να είμαστε στεναροί στο θέμα αυτό. Να μην χωρίσουμε τα πράγματα σε εξάπτυχο από τη μια μεριά και Ευρώπη 2020. Και επανέρχομαι στο ερώτημα. Δεν θα σας εκπλήξει. Το θέμα του από πού θα προέλθουν οι νέες ανταγωνιστικές δραστηριότητες. Και αυτό θα το πω με την οπτική γωνία μίας πρασίνου. Έχουμε ήδη εντοπίσει κέριους τομείς όπου μπορεί να υπάρξει μια τέτοια ανταγωνιστικότητα. Είναι η πορεία προς μια κοινωνία χαμηλής χρήσης άνθρακος και είναι η δημιουργία νέων πυρήνων βιώσιμης ανάπτυξης που μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Δεν θέλω τώρα να βάλω την κασκέτα της πράσινης και να κάνω πολιτική επιχειρηματολογία. Αλλά σίγουρα η πράσινη οικονομία είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο δυναμικό και για την εσωτερική αγορά αλλά και σε επίπεδο παγκόσμιας οικονομίας. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι αν μπορέσουμε να επενδύσουμε για να έχουμε νέα προϊόντα, να έχουμε νέες διεργασίες, να έχουμε πιο αποδοτικές δραστηριότητες. Αυτό θα δημιουργήσει περισσότερε θέσει εργασία από ένα σενάριο business as usual και θα μα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε στο σημείο αυτό, γιατί μόνο όταν γίνει σαφές ότι έχουμε κάποιε συγκεκριμένε ιδέε για το πώ θα μπορέσουμε να κάνουμε πιο ανταγωνιστική την Ευρώπη, τότε μπορούμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση αποδίδει περισσότερου καρπού από μια στενά εθνική προσέγγιση και έτσι μπορούμε να κερδίσουμε αυτή την διαμάχη. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε με ποια μορφή ο ευρωπαϊκός πολιτισμός θα βοηθήσει να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις για την ανταγωνιστικότητα. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι τώρα που υπάρχουν. Θα πρέπει να τονίσουμε γιατί είναι το κατάλληλο εργαλείο ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός το καλύτερο όχημα για τις μελλοντικέ αυτές επενδύσεις. Δεν πρέπει όμως να σημαίνει αυτό ότι τα κράτη-μέλη θα πούν εντάξει τότε εμείς δεν χρειάζεται να επενδύσουμε γιατί έτσι θα χάσουμε τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας και του 2020. Γι' αυτό στη συνδιάσκεψη της 22ης ματιού, όταν συζητήσουμε για τους κοινού μας στόχους, να τονίσουμε αυτό το πράγμα ότι δεν πρέπει να παίζουμε τους κακούς Ευρωπαίους και τους καλούς, τα, τις καλές εθνικές κυβερνήσεις. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει μια σαφήνεια στη συζήτηση μεταξύ εθνικών κοινοβουλευτικών για τον προϋπολογισμό και της ε, και της ε, Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η, η, συγγνώμη, Έλγα, όχι Ιούτα, συγγνώμη. Δίνω το λόγο μου στη Γιούτα, που δεν λέγεται Έλγα. Ευχαριστώ. Τρία πράγματα θέλω να πω. Και εγώ πιστεύω ότι οι πράσινοι θέλουν να οικειοποιηθούν την έννοια της πράσινης ανάπτυξης. Σε όλα τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου στα τελευταία δυόμιση χρόνια, όλοι πηγαίνουμε προς την ίδια κατεύθυνση και υπάρχει μια ευρεία πλειοψηφία που υποστηρίζει την πράσινη ανάπτυξη και έχουμε όλοι προσαρμοστεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Σημείο υπαριθμών 2. Το θέμα της συνεργασίας με την Κομισιόν. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κομισιόν. Θα ήθελα να πω ότι είμαι κάπως ε, ανήσυχη γιατί αυτό που είπε ο Ράιμερ ότι δεν διαθέτουμε τις ίδιες πληροφορίες όπως η Κομισιόν ή το Συμβούλιο και ότι μόνο με το να ενοχλούμε τον κόσμο και να γινόμαστε φορτικοί θα αποκομίσουμε αυτές τις πληροφορίες. Αυτό για μένα είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα και αυτό που είπε ο Ζαν Λουκ, ότι δεν έχουμε τα αριθμητικά στοιχεία για το πώς θα τροποποιηθούν οι συνεισφορές των κρατών μελών όταν ε, τροποποιήσουν τις ε, συνεισφορές τους και πρέπει να βασισόμαστε περισσότερο σε ίδιους πόρους. Όταν μιλάμε με εκπροσώπους της Κομισιόν, όταν μιλάμε με μέλη του πολιτικού γραφείου των ε, επιτρόπων, εγώ πάντα ανησυχώ όταν μας παρουσιάζουν τη συζήτηση στο Προεδρείο, τι ακριβώς έλαβε χώρα και έλεγε μετά εμείς θα κάνουμε, εμείς θα κάνουμε εκείνο, εμείς το τρίτο θα κάνουμε. Δηλαδή ουσιαστικά στο μυαλό τους υπάρχει η Κομισιόν και το Συμβούλιο, αλλά δεν υπάρχει αυτό το οποίο μας είχε υποσχεθεί ο Γιάννης Λεβαντός και ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία η Κομισιόν θα είναι ο ε, έντιμος διαμεσολαβητής μεταξύ, κοινοβουλίου, μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Δεν το δείχνουν καθόλου με τη φρασεολογία τους η τα μέλη του Γραφείου των Επιτρόπων ότι βλέπουν έτσι το ρόλο τους. Ουσιαστικά βλέπουν το ρόλο τους σαν αυτού μιας γραμματείας του Συμβουλίου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να υπογραμμίσω. Ένα δεύτερο στοιχείο θέλω να υποστηρίξω ότι εμείς δεν θα πάμε στη διαπραγμάτευση με συγκεκριμένα στοιχεία από τις επιμέρους κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αυτό αφορά όλες τις πτυχές της, ε, των μεσοπρόθεσμων ε, δημοσιονομικών προοπτικών ούτε για νομοθετήματα, ούτε για εκθέσεις πρωτοβουλίας. Και αυτό ισχύει και για μας τους ίδιους την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Αν δούμε τη γνωμοδότηση του κυρίου Γκοτμάνης, βλέπω ότι και εκεί δεν υπάρχουν κονδύλια. Είναι απλώς μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι κάτι το οποίο να γίνει εγκάρσια, να καλύψει όλες τις πολιτικές ομάδες. Και θα ήθελα <clears throat> να γίνει δεκτό από όλες τις πολιτικές ομάδες και μίλησα και με τον εκπρόσωπο του ΕΛΚ για τα θέματα αυτά και στην Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων αυτό θέλουμε να εξασφαλίσουμε δεν θα πετύχουμε όλα αυτά τα οποία θέλουμε με μια έκθεση πρωτοβουλία προφανώς, αλλά θα πρέπει και ο εισηγητή που προέρχεται από το ΕΛΚ να εξασφαλίσει να μην περιλαμβάνονται αριθμητικά στοιχεία σε αυτή την έκθεση πρωτοβουλία. να μην γίνει ένα κείμενο το οποίο θα παίζει το ρόλο μιας πυραμίδας πόντσι, λέει η Ιούτα. Δεν είναι ένα κείμενο λοιπόν το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία και να προσπαθεί να προχωρήσει σε μια διαπραγμάτευση για κονδύλια, να δοθούσουμε περισσότερα χρήματα εδώ ή εκεί. Πρέπει λοιπόν εμείς να είμαστε προσεκτικοί σε τέτοιες ε, εκθέσεις πρωτοβουλίας όπου παίρνουμε μια συγκεκριμένη θέση ότι δεν θα προκαταλάβουμε αυτά τα οποία θα ζητήσουμε για τα θέματα του προϋπολογισμού. Δεν πρέπει να ζητήσουμε κάτι το οποίο δεν θα συναρμόζεται με τα άλλα στοιχεία. Σας παρακαλώ λοιπόν να βγάλουμε τα αριθμητικά στοιχεία όταν έχουν εκθέσεις τέτοια αριθμητικά στοιχεία για την επόμενη ε, δημοσιονομική περίοδο. Ο κύριος Γκοτμάνης έχει το λόγο διότι αναφέρθηκε προσωπικά το όνομά του. Όχι μόνο να απαντήσω προς την κυρία Ιούτα Εν μέρη έχει δίκιο η Ιούτα. Είμαι αναπληρωτής και στην Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων και είμαι σκιώδης εισηγητής για τον νέο κανονισμό, τον βασικό νομοθετικό κανονισμό. Και το πρόβλημα έχει αρχίσει να αναφαίνεται όλο και περισσότερο. Σχετικά με τα αριθμητικά στοιχεία έχουμε πρόβλημα. Τι στοιχεία έχουμε σήμερα αριθμητικά. Έχουμε το 5% υποχρεώσεις, που δεν διαιρείται σε υποκεφάλαια και έχουμε επίσης και την πρόταση που έγινε πέρυσι τον Ιούνιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια πρόταση για αύξηση των υποχρεώσεων κατά 3,16%, 1,16 δηλαδή από αυτό που ζήτησαν οι πέντε χώρες για να παγώσουν τη δαπάνη το 2013. Και αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να διαιρεί, αν θέλετε, τους αριθμούς αυτούς. Δεν μιλάμε για ένα ακόμα, τρεις. μιλάμε για επιμέρους ποσά. Έχουν διαιρεθεί τα ποσά και ανάλογα κάθε επιτροπή καλύπτει έναν τομέα. Η περιφερειακή, σαν παράδειγμα, πήρε συγκεκριμένους αριθμούς, τους διέρεσε σε διαφορετικές περιοχές, υπομετάβαση περιοχές στόχου, τάδε περιοχές, ανταγωνιστικές περιοχές κτλ. Και προσπάθησε να συνεργαστεί μαζί τους. Το θέμα είναι αν αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Όταν εγώ προετοίμασα τη γνωμοδότησή μας ήμουνα σε πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί μπορεί η αριθμή να είναι λάθος, πολύ απλά και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί τελικά μου είχαν δώσει 7% μείωση για τις απόμακρες περιοχές, ενώ ήταν 4,7%. Λοιπόν, είναι απαράδεκτα και εγώ ζήτησα να μου δώσουν ένα υπογεγραμμένο έγγραφο το οποίο να εγγυάται τα στοιχεία αυτά. Μία απάντηση είναι καλή βέβαια. Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειών λέει ότι η αριθμή αυτή δεν είναι επίσημη το πρόβλημα όμως παραμένει σοβαρό, αν δει κανείς τα της Γεωργίας και ο Ζόρς τα ξέρει αυτά καλύτερα από μένα. Όλα παίζονται με αριθμούς. Και πώς θα το κάνουμε λοιπόν, πώς θα προχωρήσουμε αν δεν έχουμε τους πραγματικούς αριθμούς. Αν βγάλουμε όλους τους αριθμούς, τότε θα πρέπει να υπάρξει διαφορετικού τύπου προετοιμασία σε επίπεδο νομοθετικό από όλες τις ε, επιτροπές επί της ουσίας έτσι ώστε μετά από την απόφαση για το σύνολο του MFF τότε να μπορέσουμε να επανανσωματώσουμε τους αριθμούς, τα αριθμητικά στοιχεία. Αυτό όμως σημαίνει ότι οι επιμέρους κοινοβουλευτικές επιτροπές θα πρέπει να πάρουν ε, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να την διαιρέσουν στον δικό τους τομέα, να πάρουν το δικό τους κομμάτι και να εκφέρουν τη δική τους νομοδότηση. Λοιπόν, το θέμα είναι οι αριθμοί τους οποίους χρησιμοποιούμε, οι αριθμοί που μας έχει δώσει η Κομισιόν για τις απόμακρες περιφερειακές ζώνες. ζώνες τα ποσοστά τα οποία μπορεί να, στα οποία μπορεί να καταλήξουν, μπορεί να είναι αξιόπιστα, μπορεί να μην είναι αξιόπιστα, γιατί βασίζονται στα δεδομένα τα αριθμητικά τα οποία μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουμε άλλα. Λοιπόν, το θέμα είναι τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Ε, πρώτον, μπορούμε να ζητήσουμε να φύγουν όλα τα αριθμητικά στοιχεία, να μιλήσουμε για τις πολιτικές. Είναι ευκολότερο γιατί οι πολιτικές συνδέονται με τους αριθμούς, κυρίως με τις αναλογίες. Δεν αναφέρομαι σε απόλυτους αριθμούς, τουλάχιστον στις αναλογίες. Δεύτερον, αν θέλει κανείς να εργαστεί με τα νομοθετικά έγγραφα και να χρησιμοποιήσει τις μοναδικές υπάρχουσες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να λάβει υπόψη ότι τα ποσοστά δεν είναι αξιόπιστα, γιατί αντί για 10% αύξηση μπορεί να είναι πολύ μικρότερη. Και ένα πράγμα να προσθέσω, κάτι το οποίο είναι αρκετά σοβαρό και το είχα θέσει εκ νέου. Αν δει κανείς τον προϋπολογισμό του 2012, θα δει ποιο είναι το αποτέλεσμα της συμφωνίας ε, ε, με το Συμβούλιο, ε, με τους αριθμούς που μας επέβαλε το Συμβούλιο για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ξέρουμε ποιο είναι το έλλειμμα του προϋπολογισμού και για την Περιφερειακή Επιτροπή αλλά και για άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις πληρωμών. και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτές οι καθυστερήσεις στις πληρωμές ε, θα πρέπει να μας οδηγήσουν να αναδιορθώσουμε το δημοσιονομικό μας πρόγραμμα έτσι ώστε κάποια πράγματα να μην τα πληρώσουμε φέτος αλλά σε δύο-τρία χρόνια. Γίνεται αυτό αλλά έχουμε βρεθεί σε μια ανόητη ουσιαστικά κατάσταση γιατί σε ορισμένες κοινοβουλευτικέ επιτροπές υπάρχουν διαμαρτυρίες γιατί συνέβη αυτό το οποίο είχε πει ο Λεβαντόφσκι. Αν εφαρμόσουμε αυτά που συμφωνήσαμε το 12 για το 12 θα έχουμε πάρα πολλά ελλείμματα και στη συνοχή και στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Και πώς θα βγούμε. Πρέπει να μας ζητήσουν να βγούμε από εκεί που έχουμε πέσει πια αν συζητάει κανείς με το Συμβούλιο, ε, τους λέμε, θέλουν συνέχεια να μειώνουν, να μειώνουν, να μειώνουν, αλλά στο τέλος μένει ένα ψέμα. Ας εγκαταλείψουμε τις πολιτικές αυτές, διότι δεν είμαστε σε θέση να τις χρηματοδοτήσουμε. Το ερώτημα τίθεται λοιπόν, θα δουλέψουμε με αριθμούς ή θα δουλέψουμε χωρίς αριθμούς. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να πείσει κανείς την Περιφερειακή Επιτροπή ή την Ήτρε να δουλέψει χωρίς καθόλου αριθμητικά στοιχεία. Ούτε καν αναλογίες. Δεν είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Oui, je vous Σας ευχαριστώ, Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα απαντήσω σε όλα αυτά τα οποία λέχθηκαν. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Κοτσμάνης. Από τη μία πλευρά η Επιτροπή μας και η ομάδα επαφής επιμένουν στο γεγονός ότι αν δεν υπάρξει μια συνολική συμφωνία για τα θέματα αυτά είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μια ε, προσέγγιση και βλέπουμε ότι οι επιμέρους επιτροπές ήδη έχουν προχωρήσει με τις δικές τους προβλέψεις. Για τις επιμέρους επιτροπές υπάρχει και η δυσκολία και ο πειρασμός. Η δυσκολία είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνουν νομοθετικά κείμενα χωρίς να ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι εύκολο αυτό και υπάρχει και ο πειρασμός ο οποίος υποκρύπτεται να προχωρήσουν, να είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα διεκδικήσουν συγκεκριμένα χρήματα, συγκεκριμένα ποσά, αυτό το οποίο το ανέφερε πολύ σωστά ο κύριος Μπέργκε, να προσπαθήσουν να βγουν στην αρχή της ουράς και να βγουν από το πλαίσιο των συμπερασμάτων της Επιτροπής Σούρε. Μήπως τώρα μπορώ να κάνω μια πρόταση, γιατί δεν έχω ακούσει καμία συγκεκριμένη πρόταση για να απλοποιήσουμε τώρα το πρόβλημα αυτό. να πούμε απλώς στις επιμέρους επιτροπές προσπαθήστε να έχετε εκθέσεις νομοθετικές χωρίς στοιχεία. Εγώ δεν μπορώ να κάνω μια ελευκό έκθεση ως συζητητής Γιατί τα νομοθετικά μέτρα βασίζονται στα στοιχεία και τα στοιχεία βασίζονται στα νομοθετήματα και επομένως έχουμε μια στενή σύνδεση και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είπανε πολύ ότι ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι η πολιτική μπορεί να είναι η συνέχεια του πολέμου με άλλα μέσα. <clears throat> είναι απαραίτητο. Λοιπόν, ξέρω ότι είναι κυρίαρχες οι επιτροπές στα θέματα τις αρμοδιότητές τους. Ελπίζω ότι η ομάδα επαφής θα εξασφαλίσει τουλάχιστον οι επιμέρους θεματικές επιτροπές να καθυστερήσουν την ψήφιση των θέσεών τους για το σύνολο των προγραμμάτων μέχρι ότου η ομάδα επαφής να έχουν επαρκώς καθορίσει τη στάση τους για να επιτρέψουν στις επιτροπές να θέσουν αριθμητικά στοιχεία. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί πρέπει να πάρουν οι επιτροπές το σύνολο των αποφάσεων τους μέχρι τον ε, Ιούνιο σε συνθήκες που θα θέσουν ένα αμφιβόλο την ε, διαπραγμάτευση για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές ενώ είναι αποφάσεις οι οποίες θα εφαρμοστούν μονάχα το 2014 και επέκεινα. Εάν λοιπόν καθυστερήσουμε τις αποφάσεις των επιτροπών μέχρι μια χρονική στιγμή που θα έχουν προχωρήσει διαπραγματεύσεις, τότε θα μπορούν να ψηφίσουν για αριθμητικά στοιχεία, βάζοντας όμως σε επίπεδο συν... τα αριθμητικά αυτά στοιχεία με το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Αλλιώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε στο θέμα και ο Ράιμερ θα θέλει να κάνει διευκρινής, αλλά έχει στήσει πρώτος το λόγο Λάιον. Ευχαριστώ θα ήθελα να συνεχίσω το πνεύμα των δύο προηγούμενων παρεμβάσεων, γιατί αν πράγματι θέλουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη διαπραγματευτική άποψη, τότε το έγγραφο της ΣΟΥΡΕ θα πρέπει να γίνει δεκτό από όλους σαν το σημείο εκκίνησης. Αλλά θα πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των επιτροπών. Άμα θέλουμε να τους ζητήσουμε να προχωρήσουν στην ομοθετική τους δραστηριότητα, χρειάζονται κάποιες διαβεβαιώσεις ότι οι απόψεις τους θα γίνονται υπόψη, θα λαμβάνονται υπόψη σε θέματα τέτοιου είδους, όπως τη Γεωργία. Ένα βασικό θέμα είναι η ανακατανομή των ποσοστώσεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Στη Γεωργία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και μιλούσαν για κάποιον τρόπο τον οποίο η Επιτροπή πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η ανακατανομή Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις γύρω από αυτό, δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα. Και τίθεται λοιπόν το πώς θα αντιμετωπίσουμε αναεπιτροπή την πρόταση αυτή. Πώς θα εκφραστούμε σε σχέση με αυτόν τον τύπο ανακατανομής, τον αριθμητικό. Τελικά η απόφαση θα είναι μια πολιτική απόφαση, θα πρέπει να αποφασιστεί από το ε, Συμβούλιο. Θα δούμε τι θα γίνει τότε, αλλά θα πρέπει να πείσουμε τις κοινοβουλευτικές επιτροπές να προχωρήσουν στην ομοθετική τους δραστηριότητα σχετικά με τη δυνατότητα έκφρασης των απόψεων τους στην περίπτωση που δεν υπάρξει μια πρώτη συμφωνία στο Συμβούλιο. Για να είναι γνωστές οι απόψεις ενός από τους νομοθέτες. Ο μοναδικός τρόπος λοιπόν για να προχωρήσουμε είναι να τους διαβεβαιώσουμε ότι αν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στους τελικούς αριθμούς, τότε θα πρέπει να αντικατοπτριστούν στις απόψεις τις οποίες έχουν εκφράσει. Και να δούμε τι σημαίνει αυτό για τις αλλαγές στο συγκεκριμένο τομέα. Ράιμερ. Το τελευταίο που αναφέρθηκε τώρα δεν αποτελεί πρόβλημα. Αν οι κατευθυντήρες γραμμές ισχύσουν, θα γίνει η εργασία στην ε, Κομισιόν, θα ψηφιστούν και οι τροπολογίες και θα αναβληθεί η τελική ψηφοφορία. Επομένως δεν θα υπάρξει καμία θέση για συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, αλλά θα υπάρξει προσαρμογή η συμφωνία αυτή στην ε, ανάγκη να μην να έρθουν εγκαίρως στην ε, Ολομέλεια τα θέματα αυτά από κοινού και συγχρόνως και να μην εμποδιστεί η πρόθεση στην Ολομέλεια των θεμάτων αυτών από τη μη ψήφιση. Εμείς έχουμε συνδέσει τις προοπτικές στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ με την διατύπωση ότι αν τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να δώσουν αυτά τα χρήματα, τότε θα πρέπει να καταρτήσουν τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο, ένα κατάλογο αρνητικών προτεραιοτήτων που δεν θα υλοποιηθούν. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στους εισηγητές στις επιτροπές να έχουν μια συγκεκριμένη προσέγγιση. Λοιπόν, έχουμε τη διατύπωση της Επιτροπής Σούρε και ξέρουμε ότι η Κομισιόν μας προτείνει κάτι που είναι κάπως λιγότερο από αυτά τα οποία αναφέρει η Επιτροπή Σούρε. Αν λοιπόν δεν έχουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση για όλα αυτά τα θέματα, θα πρέπει να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να μας πει σε επίπεδο περιεχομένου ποιες είναι οι προτεραιότητες που δεν θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν. Αυτό δίνει αρκετό περιθώριο στις επιτροπές να προετοιμαστούν για μια κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αντιπαράθεση. Για ένα σημείο τώρα θέλω να σταθώ οι επιτροπές οι οποίες δεν θα ακολουθήσουν αυτούς τους κανόνες του παιχνιδιού και οι οποίες θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν εκ των προτέρων συμφωνίες με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ξέρω πώς γίνεται αυτά, προσπαθούν οι Γενικοί Διευθυντές και οι Επίτροποι να κάνουν τέτοιες συμφωνίες στο Κοινοβούλιο και αν είναι έτοιμες <clears throat> να υποστηρίξουν <clears throat> δικές τους προτάσεις θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει όχι μονάχα από τον Επίτροπο ε, για τα θέματα προϋπολογισμού αλλά και από τον πρόεδρο της Κομισιόν θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η άποψή τους και πού στέκονται για τα θέματα αυτά. Εδώ όμως θα πρέπει να έχουμε μια σαφή στάση και ως πολιτικά κόμματα, όχι να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε και τι θα κάνουμε τώρα. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε μια βασική γραμμή και αυτοί οι οποίοι δεν θα δεχτούν τη συμφωνία αυτή δεν πρέπει να τους χαϊδεύουμε στα αυτιά. Ευχαριστώ. Άλλοι έξι έχουν ζητήσει το λόγο, δεν μπορώ να τους τον δώσω. Έχουμε καθυστερήσει πολύ. Και περιμένουν οι άλλοι εισηγητές και οι εισηγήτριες. Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση, θα την ξανακάνουμε κάθε φορά στις συνεδριάσεις μας. Θέλω όμως να σας πω το εξής. Το πνεύμα αυτόν που είπε ο Ράιμερ. Πρέπει όλοι μαζί στο, είτε στο πολιετές πλαίσια, πλαίσια του πολιετούς σχεδίου είτε σε άλλες περιπτώσεις να συνεργαζόμαστε χωρίς να κάνουμε απατηλά όνειρα. Τελείωσε αυτό. τα μεγάλα και συνήθι προγράμματα εντάξει τα έχουν όλοι δεχτεί για τη γεωργία τόσα χρήματα, για τη συνοχή τόσα αλλά τα καινούργια προγράμματα είναι το θέμα. Δεν μπορούμε εκεί να ελπίζουμε συν 25% συν 50% δεν θέλουμε άλλα απατηλά όνειρα. Πρέπει να καταλήξουμε σε μία θέση όπου θα ξέρουμε ότι μπορεί να μην έχουμε παραπάνω χρήματα, μπορεί και λιγότερα και άρα χρειάζεται επιλογή. πιο περιεχόμενο θέλουμε να δώσουμε στα εγκριθέντα εγκεκριμένα προγράμματα. Θέμα αναλογίας δηλαδή, δεν είναι η απόλυτη αριθμή το θέμα. Για αυτούς έχουμε τα στοιχεία προτάσεις της Κομισιόν, τους αριθμούς για το 13 και στο τέλος η διαπραγμάτευση τι θα αλλάξει, συν 5, μείον 5% συν 10, μείον 10 κτλ. Αυτά δεν αλλάζουν την ουσία. Αντίθετα, προφανώς, αν διαπραγματευτούμε με βάση την ιδέα ότι ούτως ή άλλως στο μέλλον θα έχουμε όσα είχαμε και στο παρελθόν, τότε θα είμαστε συντηρητικοί για το περιεχόμενο των προγραμμάτων. Γιατί να αλλάξουμε μια πολιτική που ήταν ικανοποιητική μέχρι τώρα. Αν είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε τα χρήματα, τα ίδια χρήματα θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Έτσι το 20 θα καταλήξουμε στον προϋπολογισμό που χρειαζόμασταν το 90. Ενώ εγώ νομίζω ότι το 20 θα χρειαζόμαστε πολύ διαφορετικό προϋπολογισμό και μεγαλύτερο υψηλότερο δηλαδή, αλλά ακόμη και αν δεν έχει αυξηθεί πολύ, όπως προτείνει η Κομισιόν, παρόλα αυτά θα χρειάζεται πολύ διαφορετικός προϋπολογισμός από ό,τι του 90, με διαφορετικές αναλογίες. Και αυτό πρέπει να μας οθήσει να είμαστε πιο θαραλέοι στις προτάσεις που κάνουμε. Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη και η συμβουλή που σας δίνω. Σας ευχαριστώ λοιπόν, ευχαριστώ τους ηγητές. Ζητώ συγγνώμη από τις κυρίες που ζήτησαν το λόγο αλλά δεν μπόρεσαν να τον λάβουν και επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας είναι ιδιαίτερα γενές που δεν έλαβαν το λόγο. Σας προτείνω όμως τώρα να περάσουμε στο 4 την έκθεση δηλαδή του συναδέλφου Ντέρεκ Βόγγεν για τον προϋπολογισμό των άλλων οργάνων. Ορίστε, Ντερεκ. Μάλιστα, Πρόεδρε, καταρχήν να υπενθυμίσω τη διορία κατάθεσης τροπολογιών που λήγει στις 10 αύριο το πρωί. Ευχαριστώ επίσης όλους τους συναδέλφους και τις ομάδες για τη συνεργασία μας και τις συζητήσεις που κάναμε για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου το 2013. Σήμερα θα επικεντρωθώ στα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ε, συνδιαλλαγής που κάναμε με το Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Θα θυμάστε ότι στους υπολογισμούς του Προεδρείου προβλεπόταν μία αύξηση 2,996% και είχαμε πει να προσπαθήσουμε να σεβαστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο την πρόταση του Επιτρόπου και 1,9% αύξησης δηλαδή. Οι συνάδελφοι της Επιτροπής μας προσπάθησαν να το πετύχουν αυτό να παραμείνει η αύξηση στο 1,9% και στη συνάντηση αυτή έγινε δεκτή άποψη και από το Προεδρείο. Επίσης είπαμε ότι αν υπάρξουν εξοικονομήσεις για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου θα φροντίσουμε να μην μειωθεί η αποτελεσματικότητά του παρόλα αυτά. Για να υπάρξει όμως αύξηση μόνο 1,9% πρέπει να υπάρξουν εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό, δηλαδή να βρούμε 9 εκατομμύρια ευρώ τι θα τα κάνουμε και στην προκαταρκτική κοινή συνεδρίαση είπαμε να προσπαθήσουμε να, να διαγράψουμε το απόθεμα των τριών εκατομμυρίων και να παγώσουμε τα ναύλα και άλλες αποδοχές των βουλευτών πράγμα το οποίο μας οδηγεί σε περίπου 5 εκατομμύρια εξοικονομήσεις ακόμα λοιπόν μας λείπουν 4,5 εκατομμύρια στην προκαταρκτική λοιπόν συνάντηση ακούστηκαν ορισμένε ιδέες όπω το πώς θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε αυτά τα 4,5 εκατομμύρια. Μερικοί μίλησαν για αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας του Κοινοβουλίου, παραδείγματο χάρη των αντιπροσωπείε. Άλλοι είπαν να γίνουν εξοικονομήσεις περαιτέρω από τα ναύλα, όχι πάγωμα αλλά μείωση. Άλλοι μίλησαν για το συμπληρωματικό απόθεμα. Πρέπει όμως να είναι αρκετό για να μπορεί να αντιμετωπίσει ορισμένες έκτακτες περιστάσεις. Άλλοι μίλησαν για την καμπάνια πληροφόρησης, ιδιαίτερα ως προς τις εκλογές του 2014, ότι θα μπορούσαν να γίνουν εξοικονομήσεις και εκεί. Άλλοι επίσης μίλησαν για τις μεγάλες αυξήσεις που προβλέπονται για τα ιδρύματα, υπηρεσίες και ομάδες. Άλλοι για τον προϋπολογισμό της εκπροσώπησης που είναι πολύ χαμηλός. Τουλάχιστον να τον παγώσουμε αυτή τη θέση του προϋπολογισμού. Είναι μικρό το ποσό, αλλά έτσι συμβολικά Πολλές ιδέες ακούστηκαν λοιπόν από τους συναδέλφους στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ο Γενικός Γραμματέας και το Προεδρείο τώρα θα τα συνδυάσουν όλα αυτά. Την επόμενη εβδομάδα θα τα ακούσουμε, τις προτάσεις τους και θα γίνει και περαιτέρω συνάντηση της συνδιαλλαγής. Εκεί όμως την επόμενη εβδομάδα ελπίζω να μπορέσουμε να μειώσουμε όντως τον προϋπολογισμό σε αύξηση μόνο 1,9%. Μέχρι το φθινόπωρο θα καθοριστεί μια ομάδα εργασίας που να κάνει την αποτίμηση του προϋπολογισμού της λειτουργίας του Κοινοβουλίου και τις επόμενες εβδομάδες επίσης θα ακούσουμε έκθεση του Γενικού Γραμματέα που ζήτησε και από, από τον οποίο ζητήσαμε αποτίμηση των ναύλων. Πολλά λοιπόν θα γίνουν από τώρα μέχρι το φθινόπωρο. Ελπίζω τότε να είμαστε σε θέση να ταυτίσουμε ακόμη περισσότερες εξοικονομήσεις. Να μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι παγώσαμε τον προϋπολογισμό και ίσως και να τον μειώσουμε. Οι περισσότεροι εδώ στην Επιτροπή μας νομίζω συμφωνούν και τώρα και στο Προεδρείο υπάρχει συμφωνία, ιδίως για τα ναύλα να γίνουν οι περικοπές. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Το επόμενο στάδιο είναι τη Δευτέρα συνεδρίαση του Προεδρείου. Εγώ και ο εισηγητής θα είμαστε εκεί, ήμασταν εκεί μάλλον. Την Τρίτη έχουμε ε, τη συνδιαλλαγή. Εκεί δεν μπορώ να είμαι παρόν παρά στη μισή συνδιαλλαγή γιατί ταυτόχρονα έχουμε τη συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων στην οποία έχει προσκληθεί και ο κύριος Σούλτσου για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο μας απασχολεί και πρέπει να είμαι παρόν εκεί με τους εισηγητές, οπότε θα προεδρεύσει τις αντιπροσωπείες μας στη συνδιαλλαγή Ιούτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουν ζητήσει άλλοι το λόγο. Συνεπώς θα περάσουμε στο σημείο 5 τώρα, πάμε πίσω. Θα δώσω το λόγο στον Τζοβάνι Λαβία. Στην άκρα δεξιά, ο Τζοβάνι Λαβία έχει το λόγο. γλίστρισα στον εξτρεμισμό σήμερα, λαβία. Όπως γνωρίζετε όλοι, τα πιλωτικά προγράμματα και οι προπαρασκευαστικές δράσεις είναι στρατηγικά μέσα, τα οποία έχει στη διάθεσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που επιτρέπουν να ασκήσουμε μια κάποια μορφή νομοθετικής επιρροής στον προϋπολογισμό μέσω της πρότασης εφαρμογής ιδεών σε ε, πειραματικό σε εισαγωγικά στάδιο. Αν υπάρξει θετική κατάληξη, τότε οδηγούμεθα σε πραγματική γραμμή στον προϋπολογισμό. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας μεταφέρω κάποιες πρώτες ενδείξεις για τη διαδικασία την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε για τις προπαρασκευαστικές αυτές δράσεις στα πλαίσια του προϋπολογισμού για το 2013. Τα αποτελέσματα αυτά, στα οποία καταλήξαμε μέχρι τώρα, δείχνουν ότι είναι χρήσιμο να ξεκινήσει διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από τις αρκτικές φάσεις της διαδικασίας που θα οδηγήσει στην έγκριση του προϋπολογισμού 13. Γι' αυτό ακριβώς ανάλογα με αυτά τα οποία έχουν γίνει το 12, για το 12, θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας, με τη βοήθεια φυσικά όλων των συναδέλφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τη συμμετοχή όλων των εξειδικευμένων επιτροπών, μια προκαταρκτική φάση επιλογής των προγραμμάτων, τα οποία θα στείλουμε σε επίπεδο προσωρινού καταλόγου πιλωτικών δράσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εβδομάδα 23 της 4ης Ιουνίου, αυτή που ξεκινάει τις 4 Ιουνίου έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές να κάνει τη δική της αξιολόγηση για το εκτελεστό ημί, εκτελεστέο ημί συγγνώμη, των προπαρασκευαστικών αυτών δράσεων και των πιλωτικών προγραμμάτων. Οι προθεσμίες που έχουμε στη διάθεσή μας λοιπόν στο Κοινοβούλιο και σε επίπεδο μεμονωμένων επιτροπών για την κατάθεση αυτών των προπαρασκευαστικών δράσεων ορίζεται η 4η Ιουνίου. Μετά από αυτό θα, στείλουμε το, θα κλείσουμε τον κατάλογο και θα προχωρήσουμε σε αυτή την πρώτη αξιολόγηση. Η αξιολόγηση αυτή είναι για μας, θα έλεγα, ένα σημαντικό μέσο γιατί θα μας επιτρέψει να κάνουμε τις απαιτούμενες τροποποιήσεις εκεί όπου έχει καταστεί απαραίτητο, να βελτιώσουμε τις προτάσεις μας, ιδιαίτερα με το τέλος των προθεσμιών για την κατάθεση τροπολογιών για τον προπολογισμό που είναι ο μήνας Σεπτέμβριο. Θα υπάρξει χρόνος δηλαδή για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις ιδέες μας έτσι ώστε η τελική επιλογή να μας οδηγήσει σε εφαρμόσιμα προγράμματα και ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Αυτή η μέθοδος εργασίας όπως έχω ήδη πει τα τελευταία δύο χρόνια φάνηκε χρήσιμη. Γιατί πιστεύω ότι σε εποχές λιτότητας είναι απαραίτητο να μην ε, υπάρξει ε, μεγάλη διασπορά των πόρων, αλλά να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία θα προσθέσουν προστιθέμενη αξία και να μην προχωρήσουμε σε επιλογή προγραμμάτων τα οποία δεν θα είναι εφαρμόσιμα και θα μπλοκάρουν τα χρήματα που θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους. Λοιπόν, οι προθεσμίες ανακεφάλαιο είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει Βρισκόμαστε στο τέλος του πολιετούς δημοσιονομικού τετραετούς πλαισίου και υπάρχουν ορισμένοι τίτλοι οι οποίοι ε, περιορίζουν εν ε, τα προγράμματα αυτά τα προπαρασκευαστικά γιατί τα περιθώρια που έχουμε τα δημοσιονομικά είναι ελάχιστα. Θα περιοριστώ λοιπόν σε αυτή τη φάση να σας ε, παρουσιάσω τη σειρά που θα ακολουθήσουμε στα πλαίσια της διαδικασίας, περιλαμβάνεται και στο Combo News αυτό, έτσι ώστε να μπορέσετε όλοι μαζί από κοινού να παρακολουθήσετε τη διαδικασία αυτή. Υπάρχει η λεγόμενη εμπλοκή των κοινοβουλευτικών επιτροπών στην παρουσίαση των προπαρασκευαστικών δράσεων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα θέλαμε να συμμετέχουν όλες οι επιτροπές του Κοινοβουλίου που ενδιαφέρονται. Μέχρι τον Απρίλιο, μέχρι τις 23-24 Απριλίου, θα έχουμε τη δημοσίευση της δεύτερης ενδιάμεσης έκθεσης για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Και στη συνέχεια Μέχρι τις 28 Μαρτίου θα έχουμε ε, από την Επιτροπή Προϋπολογισμών προς όλες τις άλλες μεμονωμένες κοινοβουλευτικές επιτροπές τον πρώτο κατάλογο των εγκεκριμένων προγραμμάτων έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο έγγραφο το οποίο μέχρι τις 4 Ιουνίου θα πρέπει να αποστείλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να περάσει την αξιολόγηση επί της ουσίας για το εφαρμόσιμο ή όχι των προγραμμάτων. Θα μπορέσουμε λοιπόν μετά από την συλλογή των απόψεών μας και την αποστολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουμε την τελική επιλογή που θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα κατανείμουμε τον προϋπολογισμό. Αυτό που έχει σημασία είναι να χρησιμοποιήσουμε το έγγραφο το οποίο έχει στη διάθεσή μας η γραμματεία. Πρόκειται για το προσαρτημένο έγγραφο 4 και σας ζητώ να σεβαστείτε επίσης και την προθεσμία, τη χρονική, γιατί οι προτάσεις οι οποίες θα, θα παραληφθούν με καθυστέρηση δεν θα γίνουν ε, δεκτές για εξέταση. Ευχαριστώ. Η Φραντσέσκα θέλει να συμπληρώσει την παρουσία του Λαβία. Ευχαριστώ. Χαίρομαι γιατί ο Τζοβάνι Λαβία συνεχίζει να εφαρμόζει την μέθοδο, αν θέλετε, που ακολούθησε τη συνεχή εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να γλιτώσουμε χρόνο και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους. Εγώ σαν εισηγήτρια για τον προϋπολογισμό του 2012 υπογραμμίζω την μεγάλη σημασία που έχουν αυτές οι προπαρασκευαστικές δράσεις ε, του τρέχοντος έτους, που έχουμε ήδη εγκρίνει δηλαδή, και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται τα προγράμματα που επιλέξαμε πέρυσι είναι ένα βασικό σημείο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς θα προχωρήσουμε του χρόνου θα πρέπει να θέλουμε πάντα να βελτιώσουμε τη χρήση των διαθεσίμων πόρων, να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι για αυτό το ευαίσθητο πακέτο, το οποίο ε, θα έλεγα δεν είναι απλό κομματάκι του προϋπολογισμού, αλλά είναι βασικό συστατικό του. Όλα αυτά λοιπόν θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε τις κατευθύνσεις προς τις οποίες θα πρέπει να κινηθεί το Κοινοβούλιο ε, και να κάνουμε τις απαιτούμενες διορθώσεις αν αυτό αποβεί ε, πιθανό. Η κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Κάποια σχόλια επιτρέψτε μου. Ως πράσινη μπορούμε να υποστηρίξουμε τη διαδικασία η οποία έχει θεσπιστεί για τις προπαρασκευαστικές δράσεις και τα πιλωτικά προγράμματα τα τελευταία δύο χρόνια. Για την πρώτη ενδιάμεση έκθεση κομισιών λυπάμαι που δεν δόθηκαν στοιχεία για, το, για τα πιλωτικά σχέδια του EEAS. Μήπως θα μπορούσαν αυτά τα στοιχεία να συμπεριληφθούν στην επικείμενη πρόταση της Κομισιόν. Και όταν πρόκειται για την εφαρμογή και την εκτέλεση των σχεδίων αυτών, λυπάμαι που πρέπει να διαπιστώσω ότι η Γενική Διεύθυνση για τα, αγροτικά, για τα θέματα γεωργίας δεν δέχεται να εφαρμόσει προγράμματα τα οποία τα υποστηρίζουν οι πράσινοι. Αυτό είναι πραγματικά μια ε, αλαζονική αντιμετώπιση της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη έναντι των διεκδικήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζητώ λοιπόν να συμπεριφερθούν δημοκρατικά να εφαρμόσουν αυτά που ψηφίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να καταγραφεί αυτό γιατί είμαι πάρα πολύ ε, ανικανοποίητη από αυτά τα οποία έχει κάνει η Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Ευχαριστώ Χέλγα. Εμείς θα δώσουμε αυτό το μήνυμα στον Επίτροπο Τσιόλος. Εγώ προσωπικά ότι δεν, είναι, ότι δεν είναι παραδεκτό κάτι τέτοιο. Ωραία. Εάν δεν υπάρχει κάποιο άλλο ο οποίο θέλει να λάβει το λόγο, ευχαριστώ τον εισηγητή μα. Υπενθύμησε ποιον το χρονοδιάγραμμα, το έχετε στα τα κόμπου news, έτσι κι αλλιώς. Σας προτείνω να περάσουμε στο σημείο 6. 6. Να ξαναδώσω λοιπόν το λόγο στη Φραντσέσκα, διότι η απουσία σα Φραντσέσκα, έχουμε ήδη αναφερθεί στο θέμα αυτό την τελευταία φορά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να επανέλθουμε εν συντομία. Sì, molto rapidamente. Ehm, Πάρα πολύ σύντομα. Έχουμε μία πρώτη πρόταση. Όπως ε, ενθυμούνται όλοι, το θέμα αυτό ήταν ένα από τα πιο ευαίσθητα στη διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό του 2012 σχετικά με την επιπλέον συμπληρωματική χρηματοδότηση για το ΙΤΕΡ στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 12 κυρίως. Η πρόταση διορθωτική δηλαδή αφορά το 1α. Στην ουσία δεχόμαστε αυτή τη χρηματοδότηση επί της αρχής τον προϋπολογισμό αυτό για 150, 650 εκατομμύρια ευρώ αφορά και το 2013 Βέβαια είναι δημοσιονομικά ουδέτερο γιατί αντισταθμίζεται από αλλαγές που γίνονται στο 2 και στο 5. Στην ουσία λοιπόν εφαρμόζουμε με πρακτικό τρόπο στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 12 ενό τμήματος της συμφωνίας στην οποία είχαμε καταλήξει με τη συνδιαλλαγή και που αφορά άμεσα τον προϋπολογισμό του ενεστώτος έτους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη Φραντσέσκα. Η συμφωνία αυτή είναι συμβατή με την συμφωνία την οποία έχουμε κάνει και με την ερμηνεία που δίδουμε εμείς στη συμφωνία αυτή και όχι με την ερμηνεία την οποία δίδουν ορισμένα κράτη-μέλη στη συμφωνία. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Θα ήθελα να περάσουμε τώρα στο σημείο 12. Πρόκειται για τη γνωμοδότηση την οποία θα πρέπει να εκφέρουμε σαν Επιτροπή Προϋπολογισμών για τις ε, δημοσιονομικ... του φόρου για τις δημοσιονομικές συναλλαγές. Εδώ έχουμε ε, διάφορες νομικές βάσεις θα έλεγα. Στην αρχή η Επιτροπή, ο κύριος Σεμέτα, είχε προτείνει την δημιουργία ενός φόρου για τις, δημοσιονομ... για τις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που θα χρησιμεύσει σαν βάση για 27 επιμέρους εθνικούς φόρους ουσιαστικά. Εκεί αρμόδια επί της ουσίας είναι η Οικονομική Επιτροπή και εκφέρουμε γνωμοδότηση με εισηγήτρια την κυρία Γένσεν. Σε μια δεύτερη φάση θα υπάρξει ένα δεύτερο νομοθετικό κείμενο το οποίο λέγει ότι ο φόρος αυτός εφόσον ελπίζουμε κάποια στιγμή δημιουργηθεί να δοθεί στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Εκεί είμαστε εμείς η επί της ουσίας Επιτροπή και γνωμοδότρια Επιτροπή είναι η ΕΚΟΝ. Η Αν Γένσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ σύντομη θα είναι. Γιατί όπως είπατε είναι η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων που είναι η επί της ύλης αρμόδια ε, Επιτροπή και η πρόταση της Κομισιόν για ένα φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι εφικτή και μπορεί πράγματι να γίνει πραγματικότητα με τον τρόπο που προτείνει η Κομισιόν. Επομένως, από τη δική μας πλευρά και κατά την άποψή μας, αυτό το οποίο χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε είναι το κατά πόσο η πρόταση ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετους ίδιους πόρους για την ευρωπαϊκή Ένωση και αν μπορούμε να προτείνουμε στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να αντιδράσουν στο θέμα αυτό. Το δικό μου συμπέρασμα στο κείμενο της γνωμοδότησής μου είναι ότι δεδομένων των κριτηρίων που έχουμε διατυπώσει στην έκθεση Σούρε για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές θεωρούμε ότι ο φόρος αυτός χρηματοπιστωτικών συναλλαγών εκπληρεί πολλά από τα κριτήρια αυτά. Όσοι έχουν μελετήσει αυτή την πρόταση θα ξέρουν ότι δεν φορολογεί τα χρηματοπιστωτικά κέντρα, αλλά αυτούς οι οποίοι κάνουν τις συναλλαγές. Είναι λοιπόν ένας ε, επιμεριστικός νόμος, ε, επιμεριστικός συγγνώμη φόρος, και τα άλλα επιχειρήματα όπως το θέμα της ορατότητος, της επάρκειας και του μικρού κόστους ε, συλλογής. Νομίζω ότι και αυτά τα κριτήρια εκπληρούνται από ένα φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Αν λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο φόρο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εκπληρεί τα κριτήρια για ένα νέο, μια νέα πηγή ιδιών πόρων. Επομένως και εγώ ζητώ να υποστηρίξετε αυτή τη γνωμοδότηση που ζητά από την Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων να λάβει υπόψη τις ε, δύο τροποποίησεις, δύο τροπολογίες. Καταρχήν να πούμε σε μια αιτιολογική σκέψη ότι τα κονδύλια τα οποία θα συλλεγούν από τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα πρέπει να αποτελέσουν τουλάχιστον εν μέρη, αν όχι πλήρως, έσοδα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ένα τέτοιο φόρο λοιπόν θα πρέπει να είναι νέος ίδιο πόρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ένα από τα άρθρα της έκθεσης λέμε ότι τα κράτη-μέλη θα εξασφαλίσουν ότι τα ποσά τα οποία συλλέγονται από το φόρο αυτό θα μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του κανονισμού του Συμβουλίου για τους ίδιους πόρους και βάσει των διαδικασιών που θα ισχύουν. Κάνουμε λοιπόν μια αναφορά στην επόμενη εκθέση που αναφέρατε, η οποία θα έρθει στην Επιτροπή μας. Αυτά είναι λοιπόν, αυτές είναι οι δύο τροπολογίες που περιλαμβάνονται στη γνωμοδότησή μου και είναι απλά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ μπορώ να υποστηρίξω αυτά τα οποία η αν την υποστηρίζω 100% οι δύο τροπολογίες εδώ αφορούν την ε, τωρινή μας διαπραγμάτευση. Ελπίζω ότι στην πραγματικότητα θα γίνει αυτό στο Συμβούλιο, αυτό που ευχόμαστε. Ξέρουμε ότι εννέα κράτη-μέλη στις αρχές Φεβρουαρίου έστειλαν μια επιστολή στη Δανική Προεδρία ζητώντας το ταχύτερο δυνατό να υπάρξει μια θέση στην ημερήσια διάταξη του Φόρου ε, Χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ξέρω βέβαια ότι ορισμένα κράτη-μέλη πάντα θα τροχοπεδίσουν ορισμένε προσπάθειες, αλλά υπάρχουν και τα κράτη τα οποία έπανε ναι θέλουμε πράγματι να γίνει αυτή η συζήτηση για το φοροχρηματοπιστωτικό συναλλαγών και μία απόφαση του Συμβουλίου στο άμεσο μέλλον το αν θα μπορέσουν να αποτελέσουν τα, οι πρόσοδοι από αυτό το φόρο οι ίδιους πόρους, αυτό θα το δούμε. Εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρετηθούμε αυτής της ιδέας, θα πρέπει να επιμείνουμε και νομίζω ότι αυτός είναι και ο πιο σωστός δρόμος, το να αποτελέσουν ίδιο πόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Γκοτσμάνης ένα μικρό ερώτημα μονάχα και προς την ε, εισηγήτρια. Όπως ξέρουμε υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες έχουν ήδη φορολογία για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι ακριβώς φόρος των συναλλαγών, αλλά συνδέεται με το επίπεδο του ενεργητικού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Υπάρχει φορολογία στην ε, Ουγγαρία και ξέρετε ότι η Γαλλία από, από την 1η Αυγούστου θα προσπαθήσει να τέτοιο φόρο. Τι θα γίνει στο τέλος, αυτό είναι το ερώτημα, αν τα προετοιμάσουμε όλα, αν υποστηρίξουμε την Κομισιόν, θα είναι πρόσθετος αυτός ο φόρος για τις χώρες που έχουν ήδη τέτοια φορολογία ή θα αντικαταστήσει αυτούς τους φόρους που προς το παρόν εισραίουν στον εθνικό προπολογισμό. Και εδώ δεν έχω μια απάντηση. Δεν έχουν όλε οι χώρε αυτού του φόρου. Οι χώρε που δεν έχουν φόρου δεν είναι πρόβλημα τέτοιου φόρου. Αλλά εκεί που υπάρχει ήδη θεσπισμένο κάποιο φόρο αυτού του είδου, τι είδου αντίδραση μπορούμε να περιμένουμε από τι χώρε αυτέ. Αυτό δεν είναι σαφέ για μένα. Ίσως κάνουμε κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, αλλά σε τελική ανάλυση, όπως λέει η συνθήκη του Λισαβόνα θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για το θέμα αυτό. Ναι, σα ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Λαμασούρ. Απλή είναι η απάντηση. Αυτός είναι και ο στόχος της διαπραγματεύση. Αυτός είναι ο στόχος της διαπραγμάτευση. Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν φόροι, σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν φόροι. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει εδώ η δυνατότητα επίτευξης ομοφωνίας, γιατί χρειάζεται ομοφωνία για 27 χώρες, από 27 χώρες, για μια φορολογία η οποία θα είναι ε, ταυτόσιμη και στις 27 χώρες. Θα το πετύχουμε, δεν ξέρω. Ίσως να υπάρξει και εδώ ενισχυμένη συνεργασία. Πάντως, η δυνατότητα χρήσης του πόρου αυτού για την χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Προς το παρόν, αυτό το οποίο προτείνουμε είναι να υπάρξει γνωμοδότηση σαν Επιτροπή Προϋπολογισμών και πέραν αυτού τίποτα. Έτσι θα είμαστε συμβατοί και με το πνεύμα και το γράμμα της γνωμοδότησης την οποία πρέπει να δώσουμε για το περιεχόμενο της πρότασης, το ε, εύρος επιβολής, το ποσοστό επιβολής, για όλα αυτά υπεύθυνη είναι η ΕΚΟΝ. Εμείς όμως, όπως προτείνει η συγγήτρια, επιμένουμε στο ότι ο φόρος αυτός εάν δημιουργηθεί και εάν νομικά είναι δυνατό να δημιουργηθεί θα τροφοδοτήσει τον κοινοτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με αυτά τα οποία είχε προτείνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα δούμε τι θα γίνει μετά. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε πάνω σε αυτό το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα είναι να ξεκινήσουμε όντας ιδιαίτερα απεσιόδοξοι. Υπάρχει μια παροιμία στα γαλλικά, δεν ξέρω αν είναι μεταφράσιμη. Ε, το χειρότερο δεν είναι ποτέ σίγουρο. Πάντα υπάρχει ελπίδα με άλλα λόγια. Και γι' αυτό εγώ θα στοιχημάτιζα ότι θα το ε. πετύχουμε αυτό. Αλλά θα το πετύχουμε μετά από πολύ κουραστικές και μακρόχρονες διαπραγματεύσεις. Πάντως, εμείς έχουμε κάθε συμφέρον και στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής, η οποία ε, συνιστάται φυσικά ε, με πολύ μεγάλη υπομονή, η εισηγήτριά μας μας είπε ποια είναι η θέση της. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι αύριο η έκτη απογευματινή, αλλά έχει ζητήσει και άλλη μια συνάδελφος το λόγο και όπως αρνήθηκα με πολύ μεγάλη κακία να της δώσω το λόγο προηγουμένως, τον παίρνει τώρα. Ναι. Συμφωνώ με τη φρόνηση που χρειάζεται, αλλά ταυτόχρονα αισιοδοξία στη στρατηγική μας. Έχω όμως ένα ερώτημα για την εισηγήτρια. Είπαμε και φρόνηση και τόλμη. Και στη διατύπωση όταν λέμε ότι πρέπει να χρηματοδοτήσουμε συνολικά ή μερικά, αυτό είναι φρόνιμο, αλλά ερωτώ, θα το ξανασκεφτώ, δεν ξέρω αν χρειαστεί αλλαγή, αλλά θα το σκεφτώ. Μήπως δεν θα έπρεπε ήδη να πούμε ότι μιλάμε για σύνολο ή τμήμα ή μήπως δεν θα έπρεπε απλώς να πούμε να χρηματοδοτήσουμε χωρίς να βάζουμε το συνολικά ή τμηματικά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται εδώ τεράστια συζήτηση στρατηγικής, απλώς να μετρήσουμε, να δούμε πόσο τολμηροί θέλουμε να είμαστε για να δούμε πώς θα το πούμε. Κατά τα άλλα, συμφωνώ απόλυτα με τη στρατηγική που ακούστηκε. Ευχαριστούμε Ισαβέλα. Ίσως καταθέσουμε τροπολογία. Εγώ προσωπικά έχω τον πειρασμό να ακολουθήσω τη λογική που λέει ότι αρκεί να πούμε να χρηματοδοτηθεί ο προϋπολογισμός. Αυτό υπονοεί ότι θα είναι συνολικά ή μερικά. αν πούμε μόνο μερικά είναι αδύνατη διατύπωση αλλά έχω εμπιστοσύνη στην εισηγήτρια μαζί σου θα συνεννοηθείτε εκεί να βρείτε την καλύτερη διατύπωση λοιπόν οι τροπολογίες αύριο στις 18 η ώρα λίγη διωρή, 29 Μαρτίου εγκρίνεται η γνωμοδότηση η εικόν στις 24 Απριλίου Ολομέλεια τον Ιούνιο Τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο. Το 11. Προγράμματα κοινωνικής καινοτομίας. Πώς έχει αναβληθεί άψογα. Τότε πάμε στην ψηφοφορία αμέσως. αμέσως. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, Περνάμε στην ψηφοφορία πρώτον για το 16. Δεν είναι εδώ ο συνάδελφος Αλφόνση. Θα έχει όμως αντικαταστάτη. Fishing opportunities and financial contribution με τη Μοζαμβίκη. Τη συζήτηση, έντονη συζήτηση, την κάναμε την περασμένη εβδομάδα. Ψηφίζουμε λοιπόν ενιαία ψηφοφορία. Υπέρ, όχι δύο, δύο. δύο. Το πρωτόκολλο και την γνωμοδότηση. Για το πρωτόκολλο, υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Τρεις, αποχές. Το εγκρίνεται. Για την γνωμοδότηση, υπέρ. Τα χές τα ίδια. Εγκρίνεται λοιπόν με τρεις ψήφους κατά. Τώρα πάμε στο 17 έκθεση Κουνταμάνης. Γκέραν. Θα προτιμούσα να είχαμε αναβάλει την ψηφοφορία αλλά καταλαβαίνω ότι επειδή αναβλήθηκε και στη Ρέγγι ή μάλλον το αίτημα της Ρέγκη για αναβολή δεν έχει εφαρμοστεί. Υπάρχουν ακόμη αριθμοί που δεν είναι πιστικοί. Δεν είναι βέβαια και επικίνδυνοι, αλλά παρόλα αυτά, παρόλα αυτά υπάρχουν αριθμοί εδώ μέσα που και ο ίδιος ο κύριος Γκουτμάνης μας είπε ότι δεν είναι βέβαιος για αυτούς. Θα προτιμούσαμε λοιπόν αναβολή, αν όμως δεν γίνεται τότε θα ψηφίσω συστήνω στην ομάδα μου στην τελική ψηφοφορία να απόσχει λόγω των αβεβαιωτήτων αυτών. Αλλά ας μην δημιουργήσω πρόβλημα εδώ. Αν ο εισηγητής θεωρεί ότι πρέπει να ψηφίσουμε, είμαστε έτοιμοι. Αλλά τελικά θα απόσχομαι. Στο μου λένε ότι δεν έχουμε απάντηση της Επιτροπής Περίφ η οποία θα αποφασίσει στις 20 μόνο Μαρτίου όπως είχαν προβλέψει δηλαδή για την έγκριση της έκθεσης επί της ουσίας. Εμείς 21 Μαρτίου. Τι προτείνει ο εισηγητής λοιπόν ο κύριος Γκοντμάνης. Να σας εξηγήσω. Κατανοώ αυτά που ακούστηκαν γιατί και εγώ ανησύχησα όταν είδα ότι πρέπει να συνδυάσω τρεις συμβιβασμούς αλλά η αριθμοί εδώ είναι απολύτως εγκεκριμένη από την περίφ. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του κυρίου Σούριανς και των άλλων. Η αριθμή αυτή είναι εγκεκριμένη. Άλλο, δεύτερον. Είπαμε, ή θα γνωμοδοτήσουμε με τους υπάρχοντες αριθμούς, που βρίσκονται στην έκθεση της ΠΕΡΙΦ και επειδή είμαι αναπληρωτής εκεί είδα πως το συζητούν εκεί. Είναι πολύ ανήσυχοι διότι ήδη υπάρχουν περικοπές και η Κομισιόν δεν έχει απαντήσει κλπ. Εγώ προσπάθησα εδώ στην κρομοδότησή μας να βάλω ουδέτερα πράγματα Πήραμε την πρόταση της Κομισιόν, είπαμε ότι διαφωνούμε αλλά δεν επιμένουμε να υπάρξουν τα ίδια ποσά όπως πριν γιατί λένε ότι δεν είναι ρεαλιστικό αυτό και μιλάνε για περισσότερη ευελιξία. Έτσι λέει και στην έκθεση της Περίφ. Προσπάθησα λοιπόν και από ό,τι κατάλαβα επειδή αντιδρούν στους αριθμούς της Κομισιόν εμείς είπαμε ότι δεν επιμένουμε στην επαναφορά του αρχικού ποσού. Είπαμε ότι δεν πρόκειται για περικοπές μόνο στις απομακρυσμένες περιοχές αλλά παντού και στις περιοχές σύγκλησης. Και γι' αυτόν τον λόγο οι πολιτικές ομάδες θα αποφασίσουν. Εγώ όμως σας ε, ξαναλέω ότι δεν πρόκειται να βελτιωθούν τα πράγματα. Προσπάθησα να χρησιμοποιήσω πραγματικούς αριθμούς χωρίς να επιμένουμε να λέμε περισσότερα στις απομακρυσμένες κλπ. Αυτά είχα να σας πω. Γκέραν, απαντάει αυτό στην ανησυχία σου. Είσαι έτοιμος να ψηφίσεις σήμερα. Μάλιστα, μάλιστα. Αν δεν υπάρχει άλλη αντίρρηση επί του ίδιου θέματος, περνάμε στην ψηφοφορία του. Υπάρχουν πολλοί συμβιβασμοί. Έχετε όλοι τον κατάλογο ψηφοφορίας. Συμβιβασμός γάμα υπέρ. Ευχαριστώ κατά χες, χες. Ευχαριστώ εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο συμβιβασμό α υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές εγκρίνεται παρά την αντίρρηση τεσσάρων μελών. Τροπολογία 7 της σοσιαλιστικής ομάδας. Ο εισηγητής είναι κατά υπέρ. Η κατά. Οι υπόλοιποι απαρρίπτεται. Το 8 των ιδίων. Ψυχητής επίσης κατά. Υπέρ. 20 ληστέ. Και ο κύριος Χάγκλουντ. Κατά. Όλοι οι υπόλοιποι. Εκτός από τον κύριο Χάγκλουντ. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Λάσλο Σουριάνου. Εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Τα ΑΛΦΑ Έχετε κάρτες. Για να γελάσουμε λίγο τώρα με τα σκάρτας. Να ζεσταθούν και οι μηχανές. Αρχίζει η ψηφοφορία. Άμα λείπουν κάρτες να μου το πείτε. Δεν έχετε κάρτα Φραγκίσκη να μας το πείτε στο τέλος. Λοιπόν, Α, έληξε η ψηφοφορία. Έληξε. 16 υπέρ, 11 κατά. Καμία αποχή. Φραγκίσκη, πώς θα ψήφιζες. Κατά. 16-12. Εγκρίνεται. 10. Πώς, πώς. Α. 10. Συγητής κατά. κατά. Υπέρ, υπέρ. 10, ε. 10 τις κατά. Κατά. Εγκρίνεται. 11. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. χέ Εγκουρίνεται. Συμβιβασμός Β. Υπέρ. Κατά. Μάλιστα. Νομίζω οι περισσότεροι ήταν υπέρ, αλλά ας χρησιμοποιήσουμε τα σμηχανάς. Α, ψηφίσω κι εγώ, είναι λίγοι στο ΕΛΚ. Λοιπόν, έληξε. 18 υπέρ, 9 και 1 κατά, υπέρ, εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν τώρα στην τροπολογία 15 εισηγητής κατά υπέρ κατά χες εγκρίνεται Ό! όχι, όχι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Απορρίπτεται εννοούσα. 16. Ο συγκητής είναι υπέρ. Κατά. Yes, εγκρίνεται. 17. Ο συγκητής είναι κατά. Υπέρ δύο Κατά περισσότεροι. Απορρίπτεται. 17, 18 του ιδίου υπέρ. Συγκρίνεται καλά. Κατά. Αποχέ. απορρίπτεται. Αφού έχουμε τις μηχανές να κάνουμε την τελική ψηφοφορία με τη μηχανή. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται, άρχεται, άρχεται, έληξε. 18 υπέρ, 4 κατά, 5 αποχές. 6 αποχές μάλιστα. 6 αποχές γιατί είναι και η Φραγκίσκη. Εγκρίνεται, συγχαίρουμε τον κύριο Κουνταμάνη. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στις μεταφορές. Η Φραγκίσκη δεν έχει μεταφορά. You have no transfer. Δυστυχώς. Λοιπόν, μεταφορά προϋπολογισμού των άλλων οργάνων. Κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι μια τροποποίηση. Όπως παρουσιαστήκε αυτές οι προτάσεις, υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι οι οποίοι μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο ώστε στο διάστημα αυτό να διαλύσουμε κάποιες παρεξηγήσεις, να έχουμε μια καλύτερη παρουσία στον απόψεων και νομίζω ότι στις 20 Μαρτίου μπορούμε να κάνουμε την ψηφοφορία. Δεν μπορούμε βέβαια να υπερβούμε την 20 Μαρτίου. Πρόκειται για μια τροποποίηση για 2 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για το κτίριο CAD στο Λουξεμβούργο, αλλά υπάρχει ήδη μια καθυστέρηση για αυτήν την ε, ενέργεια και είναι μια μεταφορά πιστώσεων που έχει σε στόχο <clears throat> την συντήρηση των κτηρίων στις Βρυξέλλες. Είναι μια απόφαση που είχε ληφθεί ήδη από το Μάρτιο του 2010 και συμφωνήσαμε να υπάρξει αυτή η συντήρηση, αλλά υπάρχουν, ε, υπάρχει πρόσθετο κόστος που έχει δημιουργηθεί και υπάρχουν και προβλήματα ασφάλειας τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Υπήρξαν λοιπόν κάποιες αμφιβολίες σε αυτή την γνωμοδότηση, ακόμα και αν η γραμματεία μας έχει πληροφόρηση καλά για τα θέματα αυτά. Δεν μας λέει όμως ακόμα η γραμματεία του Κοινοβουλίου αν πρόκειται για όλα τα κτίρια ή πρόκειται μονάχα για ορισμένα κτίρια που έχουν αυξημένες ανάγκες και επομένως υπάρχει το ερώτημα του κατά πόσο αυτή η συντήρηση αφορά όλα τα κτίρια των Βρυξελών. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποιος αρμόδιος ο οποίος θα μπορούσε να μας απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Σας ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος, Ο Ντέρεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Μόλις χθες πήρα την έκθεση αυτή και δεν ήταν ούτε στα αγγλικά ούτε στα ουαλικά η άλλη γοηδελική έκφραση. Δεν μπορούσα λοιπόν να τα μελετήσω και μπορούμε επομένω να ακολουθήσουμε και την πρόταση του εισηγητή να αναβάλουμε την ψηφοφορία μέχρι τις 20 και έτσι θα έχουν όλη την ευκαιρία να δουν αν θέλουν να κάνουν κάποια σχόλια και να τροποποιήσουν τη θέση τους. Ευχαριστώ πολύ. Για το θέμα αυτό δεν θα ψηφίσουμε σήμερα. Θα δώσουμε το χρόνο στο χρόνο για να κάνουμε τους ε, αραβικούς χαρακτήρες για τα αριθμητικά στοιχεία να τα μεταφράσουμε στα ουαλικά, λέει ο πρόεδρος. Τούτου λεχθέντος. Έχει θέσει ερωτήματα ο εισηγητή στην αρμόδια γενική διεύθυνση, η οποία εκπροσωπείται εδώ από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση ε, Υποδομών και Επιμελητίας και μου ζητήσανε να δώσω κάποιες ε, πληροφορίες σε σχέση με την αίτηση μεταφοράς πιστώσεων. Πρόκειται για μια νέα ε, συμφωνία, ένα νέο συμβόλαιο για την ε, ανακαίνιση και συντήρηση των κτίριων στις Βρυξέλλες που θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Απρίλιο. Πρόκειται για όλα τα κτίρια όπως είπε, όπως είπε και ο εισηγητής όλα τα κτίρια των Βρυξελών, τα οποία θα καλύπτονται από αυτή τη συνθήκη, την Συμφωνία Συντήρησης. Αυτό είναι η υλοποίηση της απόφασης του Προεδρείου για το που ελήφθη το 2010. 20 χρόνια έχουμε αυτά τα κτίρια. 20 χρόνια. Και αρχίζουν να γερνάνε αυτά τα κτίρια μετά από 20 χρόνια. Γνωρίζετε επίση ότι υπήρξε και αυτό το πρόβλημα στο Στασβούργο, όπου έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι μας. Γι' αυτό έχουμε συνάψει αυτή τη σύμβαση μέσα στα πλαίσια μιας νέας πολιτικής κτίριων. Ε, πήραμε την ε, γνώμη και τις συμβουλές εμπειρογνωμόνων και έχουμε κάνει μια προκήρυξη για μια νέα α, σύμβαση συντήρησης, η οποία βέβαια θα είναι πιο πολυδάπανη από ό,τι στο παρελθόν, αλλά πρέπει να δώσουμε τα απαραίτητα κονδύλια. Είναι απαραίτητο να υπάρξει λοιπόν η συντήρηση <clears throat> των ε, εγκαταστάσεων στα περισσότερα κτίρια. Χρειάζεται να ελέγξουμε και να ανακαινήσουμε τις ε, εγκαταστάσεις κλιματισμού, ηλεκτροδότησης, ε, θέρμανσης. θα πρέπει να ελεγχθούν όλες οι εγκαταστάσεις και επίσης φυσικά θα πρέπει να υπάρξει και μια καθημερινή παρακολούθηση όλων των εγκαταστάσεων. Και η σύμβαση αυτή μας δίνει μια πλήρη εγγύηση, δηλαδή είμαστε απόλυτα εξασφαλισμένοι έναντι οποιοδήποτε κόστους επισκευής το οποίο θα προκύψει. Όταν τώρα δεν ε, χρησιμοποιηθεί αυτός ο προϋπολογισμός ο οποίος προβλέπεται, τότε το Κοινοβούλιο θα πάρει το υπόλοιπο πίσω. Αλλά άμα ξεπεράσει αυτό το επίπεδο του προϋπολογισμού το κόστος της επισκευής, τότε είναι η εταιρεία, η ανάδοχος η οποία πρέπει να πληρώσει το πρόσθετο κόστος. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρχει και περισσότερο προσωπικό το οποίο θα παρακολουθεί τα κτίρια και έχει ανέλθει το επίπεδο των προσόντων των ε, ατόμων αυτό και ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε μία σειρά από τεθειμένους στόχους και για κάθε στόχο υπάρχει μία σειρά δικτών που καθορίζουν πότε θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση του αναδο, της ανάδοχης εταιρεία για να κάνει τις ε, επισκευές. Αν δεν επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, παραγωγός χάρη για τη διαθεσιμότητα των κτηρίων και των ε, υποδομών, πρέπει η ανάδοχος εταιρεία να πληρώσει κάποιο πρόστιμο. Το ίδιο αναφέρεται και σε σχέση με την ποιότητα του αέρος στις ε, αίθουσες. Όλα αυτά καλύπτουν τις ε, προδιαγραφές για το περιβάλλον, για την εξοικονόμηση ενέργειας κτλ. Αυτά λοιπόν καταρχήν τα πιο σημαντικά θέματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμού να δούμε όλες τις επιμέρους διατάξεις. Σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις προφορικές εξηγήσεις. Ο εισηγητής μας θα εξετάσει το λεπτομερές κείμενο και θα με συνημερώσει την επόμενη φορά έτσι ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε γνωρίζοντας περί τίνος πρόκειται. Η Μόνικα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία, εγώ νομίζω ότι πράγματι έχει νόημα στον τομέα της ανακαίνησης και της ε, συντήρηση των κτηρίων είναι πολύ καλό που βρήκαμε μία συστηματική λύση. Είναι καλύτερο να διατηρούμε τα κτίρια σε καλή κατάσταση γιατί μετά τα μερεμέτια κοστίζουν πάντα περισσότερο. Έχω και κάποια ερωτήματα σε σχέση με την διαδικασία αυτή ε, διαγωνισμού που ακολουθήθηκε. <coughs> <coughs> θα ήθελα να ξέρω και τις λεπτομέρειε, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα καταλήξουμε σε μια θετική ψηφοφορία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και σήμερα να ψηφίσω μετά από τις εξηγήσεις που έχουν δοθεί από την, ε, τις του Κοινοβουλίου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Φυσικά να ψηφίσουμε ούτε και στις 20 Μαρτίου. Εγώ φυσικά οικοθενοείτε ότι σας ζητώ τη θετική σας ψήφο για αυτή την τροποποίηση. Ωραία, τρέμπιαν λέει ο πρόεδρο. Καλώς, με την επιφύλαξη βέβαια των γνωμοδοτήσεων, τις οποίες μέχρι τότε θα μας στείλουν οι συνάδελφοι ή θα μπορούσαν να στείλουν. Ένα τελευταίο θέμα, το οποίο μπορεί να χρειαστεί να ψηφίσουμε, είναι η πολιτική ε, για τα κτίρια. Buildings policy, λέει ο πρόεδρο έχει καμία σχέση η πρόταση αυτή με τον τέος Ούγκρο Πρωθυπουργό Χόρβατ. <laughs> Εδώ έχουμε μόνο θετικά στοιχεία. Καλά. Έχουμε πάρει πάρα πολύ πρόσφατα τα στοιχεία της Κομισιόν για τα δύο σχέδια κτηριακού χαρακτήρα Γι' αυτό είμαι υποχρεωμένη να σας πω στην αρχή ότι με κάποια με, κάποια, με κάποιο ενδιαφέρον είδα ότι διαφέρει πάρα πολύ η έννοια του κατεπήγοντος για το Κοινοβούλιο και για την Κομισιόν αλλά αυτό το οποίο η Κομισιόν έχει κάνει είναι εμπεριστατωμένο μου έχει δώσει μονάχα τρει μέρε για να αντιδράσω. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τα θέματα αυτά. Νομίζω και τα δύο σχέδια μπορούν να υποστηριχθούν. Πρόκειται για δύο κτίρια. Το κτίριο Όρπαν και το COV4. Θα υπάρξουν λοιπόν συμβάσεις εξυπηρέτησης μέσα στα πλαίσια των κτηρίων αυτών Έχουμε το κτίριο STM, το οποίο όμως είναι ιδιαίτερα πολυδάπανο και με τη νέα συμφωνία θα εξοικονομήσουμε 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. Έχουμε 39.000 ε, τετραγωνικά μέτρα για γραφεία και τα οποία θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες περίπου χιλίων ατόμων. 307 ε, ευρώ το τετραγωνικό είναι το κόστος ε, ε, ενοικίασης και περίπου 600.000 είναι το κόστος για την ενεργειακή υποστήριξη των κτηρίων, 400.000 περίπου για την ασφάλεια και ελπίζουμε μέχρι το Δεκέμβριο του 2011 θα έχει κλείσει η σύμβαση αυτή και θα μπορούμε επομένως να 12 όχι 11, να εγκατασταθούμε στο κτίριο αυτό. Φυσικά είναι απαραίτητο να γίνουν οι απαραίτητες ε, συμφωνίες με τις εταιρείες και να καταλήξουμε και στις ε, ρήτρες που είχαμε ζητήσει εμείς. Το σχέδιο Orban έχει περίπου 24 και μισό χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, 55.000 μαζί με το πάρκινγκ και υπάρχει και χώρος για παρκάρισμα ε, ποδηλάτων, 150 ποδηλάτων. Η κατάσταση του κτηρίου είναι καινούριο, είναι σε πάρα πολύ καλή ε, θέση, είναι εύκολα προσβάσιμο από το κοινοβούλιο, θέλει 2-3 λεπτά περπάτημα μονάχα και δεν έχουμε προβλήματα με αμίαντο ή οτιδήποτε τέτοιο γιατί είναι ένα καινούριο κτίριο και έχουμε περίοδο ενοικίασης 20 χρόνια, 25, 23 χρόνια μάλλον. Θα έχουμε τώρα περίπου 10 τετραγωνικά μέτρα για κάθε άτομο. Και δεν έχουμε ακόμα ε, δεν έχουμε κάποιες ε, προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Θα έχουμε μια συνολική οικονομία 3,9 εκατομμυρίων για 23 ε, μήνες. Και μετά θα περάσει σε ένα άλλο επίπεδο η τιμή ανά τετραγωνικό Όλα αυτά λοιπόν μας έρχονται πολύ πιο φτηνά από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ πιο θετικές οι συνθήκες λοιπόν για το κόστος και αν υπολογίσουμε ότι θα χρειαστούμε και το κόστος επισκευής και ανακαίνησης που είναι περίπου 7 ευρώ τετραγωνικό έχουμε ακόμα ένα συνολικό κόστος 17.000 ανά τετραγωνικό. Θα έχουμε περισσότερο χώρο στη διάθεσή μας εξάλλου, περίπου 20.000 τετραγωνικά. Υπάρχουν καντίνες κτλ. 20 χρόνια θα έχουμε την χρήση κτησία και υπάρχει και μία αν θέλαμε να έχουμε μία ρήτρα για πρόορη διακοπή του συμβολέου, θα κόστιζε περισσότερο. Έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε 560 άτομα στο χώρο αυτό και υπήρξαν πραγματικά οι συνθήκες κατεπήγοντος. Η βελγική κυβέρνηση είχε ζητήσει είχε έρθει σε μια σύγκρουση με την Κομισιόν για ένα κτίριο το οποίο ήθελε να διεκδικήσει και η Κομισιόν. Και τελικά αυτό κατέληξε στα χέρια του βελγικού ε, κράτους 3,87 θα είναι το κτίριο αυτό. 24 μήνες δεν θα έχει τα βασικά τέλη να καταβάλει το Κοινοβούλιο και έτσι οι συνθήκες για την παροχή των κτιρίων αυτών είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. 160 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο θα κοστίσει και αν βγάλουμε το γεγονός ότι έχουμε επί 24 μήνες δεν πρέπει να πληρώνουμε τέλη, αυτό θα είναι πάρα πολύ θετικό. Το, ο εξοπλισμός του κτηρίου θα γίνει στα επόμενα αν αποσβεστεί σε 15 χρόνια θα μειωθεί το πραγματικό κόστος και γι' αυτό θέλουμε να υποστηρίξουμε την Κομισιόν περιπτώσει και τα δύο κτίρια είναι πολύ καλά. Έχει υπάρξει πολύ καλός προγραμματισμός και παρά την οκίτητα έχουμε καταφέρει να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα της Κομισιόν μέσα στα πλαίσια της αγοράς κτίριων. Και σας ζητώ λοιπόν να υποστηρίξετε. Συγγνώμη που τα είπα τόσο γρήγορα όλα αυτά τα αριθμιστικά στοιχεία. Ε, όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Από ό,τι κατάλαβα όμως από αυτά που είπατε, Πιστεύετε ότι τα δύο αυτά, οι δύο αυτές προτάσεις είναι αποδεκτές. Και δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι συγκεκριμένο. Συνεχίζει χωρίς μικρόφωνο ο πρόεδρος, δεν τον ακούμε. Λοιπόν, ε, θεωρεί η συγγήτρια ότι είναι καλά τα προγράμματα αυτά, τα σχέδια αυτά και δεν, ε, δεν προτείνει να υπάρξει γνωμοδότηση. Πριν κλείσουμε, θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο λέγοντας ότι προηγουμένως δεν είχαμε χρόνο. Λοιπόν, η Ντεβ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θέλω να κάνω ένα επίσημο παράπονο γιατί δεν είχα δυνατότητα να μιλήσω αλλά τώρα εσείς μου δώσατε αυτή τη δυνατότητα οπότε αποσύρω τη διαμαρτυρία μου. Έχει κλείσει η συζήτηση και είναι δύσκολο να επανέλθω εκεί που βρισκόμαστε στο παρελθόν. Αλλά η συζήτηση για το χρηματοδοτικό πλαίσιο που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια σωστή στρατηγική σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι συζητάμε πάρα πολύ για, το, για τη διαδικασία και δεν συζητάμε αρκετά για το περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή γίνονται πράγματα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Έχουμε ειδήσει από το Συμβούλιο για το Ταμείο Συνοχής. Ξέρουμε ότι κάποια σχέδια κινδυνεύουν να παραλύσουν με το, <clears throat> με το πρόσχημα νομικών προβλημάτων. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Έχουμε ένα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα με τις πληρωμές. Ε, μόνο στο Ταμείο Συνοχής μπορούν να γίνουν περικοπές στις πιστώσεις υποχρεώσεων. Πρέπει λοιπόν να είμαστε καλύτερα πληροφορημένοι για αυτά τα οποία ζητάει η Κομισιόν. Μας στέλνει ορισμένα δημοσιονομικά δελτία. Καλό είναι αυτό, αλλά αυτό με τον οποίο πρέπει να διαπραγματευτούμε είναι το Συμβούλιο και το Συμβούλιο έχει πολλά προβλήματα για να μπορέσουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία μεταξύ του, μεταξύ των αναγκών υποστήριξη τη συνοχή και υποστήριξη τη λιτότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλα αυτά τα στοιχεία, να δούμε πώ προχωρούν οι διαπραγματεύσει στου κόλπου του Συμβουλίου και να έχουμε περισσότερη ουσία και όχι μονάχα να λειτουργούμε με τα δημοσιονομικά δελτία. Διαμαρτυρόμαστε ότι δεν έχουμε πληροφορίες, αλλά τις λίγες πληροφορίες που έχουμε δεν τις έχουμε διαξέλθει, όπως αυτά σε δημοσιονομικά δελτία. Πάρα πολύ συζητήσαμε λοιπόν για το στρατηγικό και το, προσε... το διαδικαστικό, αλλά όχι για την ουσία της διαπραγματεύσεως και αυτό το οποίο αρχίζει να έρχεται από την Κομισιόν και το Συμβούλιο για τις προτάσεις αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ, Άιντα. Στην ουσία όμως η διαπραγμάτευση δεν ξεκίνησε. Δεν έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση ούτε στο Συμβούλιο ούτε ανάμεσα στο Συμβούλιο και σε εμά. Και δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν από το Συμβούλιο του Ιουνίου. Προς το παρόν, οι θέσεις και οι προτάσεις για το χρονοδιάγραμμα εργασίας των Δανών της Προεδρίας της Δανικής προβλέπει ότι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του μηνός Μαΐου θα ασχοληθεί θα εξετάσει με το λεγόμενο negotiating box, το κοιτίον διαπραγμάτευσης, το οποίο δεν θα περιλαμβάνει όμως κανένα αριθμητικό στοιχείο και θα είναι μια απλή ανακεφαλαίωση των θέσεων των 27 αντιπροσωπιών και της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και υποθέτω ότι το συμπέρασμα θα είναι να προσκληθεί το Συμβούλιο στο να συζητήσει κάποια γενικότερα θέματα και κάποιους απλούς προσανατολισμούς. Αυτό θα υποβληθεί στη συνάντηση κορυφής του Ιουνίου για να γίνει αντικείμενο μιας πρώτης συζήτησης. Και επί τη βάση αυτής της πρώτης συζήτησης θα γνωρίζουμε αν μπορεί να ξεκινήσει η πραγματική διαπραγμάτευση για τους αριθμούς ή εάν το Συμβούλιο το ίδιο έχει περισσότερο χρόνο, θέλει περισσότερο χρόνο. Αυτό που μας καθυστερεί είναι το θέμα της κρίσης του χρέους και της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών, σε επίπεδο συνάντησης Υπουργών Οικονομικών ασχολούνται αποκλειστικά με το θέμα της Ελλάδας και με το να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για το για το Fiscal Compact. Θα ξεκινήσουν τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό 14 με 20 μετά τον Ιούνιο, το ενωρίτερο. Η δυσκολία για μας είναι ότι θα πρέπει να υποφεληθούμε από την περίοδο που μεσολαβεί έτσι ώστε να οργανώσουμε σωστά τη μέθοδο εργασία μας, να διευκρινίσουμε καλά τις στρατηγικές μας και να αξιολογήσουμε το συσχετισμό δυνάμεων στο αντίπαλο μέρος. Και η συνάντηση της 22ης Μαρτίου θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί κατά τη διάρκεια της συνάντησης της διακοινοβουλευτικής που έγινε εδώ και λίγες μέρες δεν ήταν εκεί οι κυβερνήσεις μια συνάντηση που οργανώσαμε με τους συναδέλφους των Επιτροπών Απασχόλησης και της Οικονομικής Επιτροπής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το θέμα ήταν οι εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές, αλλά ήδη υπήρξε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων ενδιαφέρουσα, όπως ακούστηκε πριν. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και άλλη ευκαιρία για να κατανοήσουμε περισσότερο το τι πιστεύουν και οι άλλοι. Χτες και προχτές ήμουνα στο Βερολίνο. Είχα κάποιες επαφές με τους Γερμανούς. Είναι σαφές ότι και στο Παρίσι και στο Βερολίνο αναγνωρίζουν το ότι θα πρέπει να υπάρξει διαπραγμάτευση για το πολιετές πλαίσιο, αλλά δεν έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους εκτός από αυτό που λέει ότι όσο μικρότερος είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός τόσο το καλύτερο γιατί μειώνεται η εθνική συνεισφορά. Ε, τώρα αυτό δεν είναι και θέση διαπραγμάτευσης, είναι θέση αναμονής. Προς το παρόν λοιπόν η άμεση οι άμεσες συνέπειες της κρίσης απασχολούν όλο τον κόσμο. Αυτή στιγμή αυτό το χρηματοπιστωτικό Φουκουσίμα αρχίσει να ψύχεται, τότε θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Και αυτό που είπε η Ειντερ έχει δίκιο απολύτως. Λοιπόν, αυτά συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Επόμενη συνάντηση την 21η Μαρτίου στις 9 το πρωί και το μεσημέρι μετά. Τέλος.